Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσει η συνεδρίασή μας. Sur euh, l'adoption Ως προς την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σα επισημάνω κάποιες αλλαγές για την απογευματινή μας και την αυριανή μας συνεδρίαση. Ο Επίτροπος Σαλμούνια, που κανονικά θα ερχόταν στις 3 και 4, μου ζήτησε να έρθει αργότερα, κατά τις 5. Και φυσικά συμφώνησα. Οπότε το σημείο 4 της ημέρησης διάταξης θα αρχίσει στις 5 και όχι στις 3 και 4. Θα προηγηθεί εξέταση του σημείου 6, αν δεν έχει αντίρρηση η συγγήτρια, η κυρία Κίνκα Γκέντς, με θέμα το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων και το Progress και το σημείο 8 για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Γνωμοδότηση της κυρίας Χάρκιν. Αυτά θα προηγηθούν τη συζήτηση με τον Επίτροπο Αλμόνια. Τώρα, από την αυριανή μέρη διάταξη, η Επιτροπή Προπολογισμών μα ζήτησε να αναβάλουμε την ψηφοφορία τη έκθεση King Guns για τι μικροχρηματοδοτήσει, προκειμένου να προλάβει η Επιτροπή Προπολογισμών να υποβάλει τη γνωμοδότησή της, κάτι που δεχτήκαμε. Οπότε, η ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού για το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για το 2010 θα γίνει πριν ε, τα σημεία 9 και 10 για τους μικροχρηματοδοτήσεις και το progress. Εδώ παρακαλώ δώστε λίγη προσοχή, γιατί ανάλογα με την ψηφοφορία που θα γίνει για τα σημεία 9 και 10, ίσως ε, ψηφίσουμε μία πρόταση ψηφίσματος για την επιτροπολογία. Και μάλιστα αν δεχτούμε την πρόταση συγκήτριας ε, να απορρίψουμε δηλαδή το μηχανισμό χρηματοδοτήσεων ε, την ε, χρηματοδότηση μάλλον του μηχανισμού χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα Progress, τότε θα έρθουμε σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η σύσταση της εισηγήτριας. Ε, οπότε σε τέτοια περίπτωση θα αντιταχθούμε σε ένα μέτρο επιτροπολογίας που εφαρμόζει το κοινοτικό πρόγραμμα Progress χωρίς να περιμένει την απόφαση και την ψηφοφορία της δικής μας Επιτροπής. Τέλος, στο σημείο 15. Προφορική ερώτηση για τη μετακατάσταση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και για την προφορική αυτή η ερώτηση για να περιληφθεί στη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου. Όταν λοιπόν ψηφίσουμε για την υπόθεση Dell της Ιρλανδίας μετά το 15 θα ψηφίσουμε και για τη μετεκατάσταση, γιατί είναι λένε τα δύο θέματα, τη ΔΕΛ και τη μετεκατάστασης. Συμφωνείτε με αυτές τι αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη. Πολύ ωραία. Και παίρνουμε στο σημείο 2, την έγκριση των πρακτικών. Δεν έχω λάβει ιδιαίτερα αιτήματα για τα πρακτικά, οπότε εγκρίνονται. Ανακοινώσει της Προέδρου. Ο συνήθως ε, η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω του web ναι. streaming. Δηλαδή υπάρχει αναμετάδοσή της μέσω του διαδικτύου. Έχετε λάβει και την ανακοίνωση που ανέκριναν οι συντονιστές σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της εξαγωγής ψηφοφορίας στην Επιτροπή μας, ώστε να εργαζόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 5 της ημέρησης διάταξης που προβλέπει την ψηφοφορία επί δύο επιστολών για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Στο Βέλγιο για τη βιομηχανία της ε, κλωστοϊφαντουργίας και στη Ιρλανδία για την επιχείρηση Dell. Μάλιστα στην Ολομέλεια συζητήσαμε αυτά τα δύο θέματα, τις δύο επιχειρήσεις. Ήδη για το Βέλγιο υπήρξε συνένεση. Για την Ιρλανδική περίπτωση, της Dell δηλαδή, θα θυμάστε ότι είχαμε υποβάλει το θέμα στους αρμόδιους επιτρόπους ανταγωνισμού και κοινωνικών υποθέσεων ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις για την υπόθεση Dell. Και σας έχουμε μοιράσει τις απαντήσεις των Επιτρόπων στα γαλλικά. Για να δείτε περί τίνος πρόκειται. Η επιστολή αυτή ως προς την ουσία δεν φωτίζει ιδιαίτερα. Απλώς υπενθυμίζει ότι στην περίπτωση αίτησης κρατικών ενισχύσεων από πλευράς Πολωνίας η στρατηγική της ΔΕΛ φάνηκε ως στρατηγική εγκατάστασης δεύτερου εργοστασίου στην Ιρλανδία και όχι με μετεγκατάσταση στην Ευρώπη. Βέβαια, κανένας δεν θέλησε να αμφισβητήσει την ενίσχυση που είχε υποσχεθεί το κράτος στους Ιρλανδούς εργαζόμενους. Σας προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε την επιστολή. Μετά την χθεσινή τροποποίηση που έγινε και από την ομάδα εργασίας στην Αρμόδια, ζητήσαμε το ΕΛΚ ζήτησε ψηφοφορία κατά τμήματα για ένα τμήμα της τροπολογίας που είχε υποβάλει η Γκουε. Αλλά το μεταξύ η ΓΚΟΕ απέσυρε αυτό το εδάφιο της τροπολογίας. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Μπορούμε να ψηφίσουμε ολόκληρη την επιστολή προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θέλει κανείς το λόγο, η κυρία Μόγα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι προσωπικώς εκπροσωπώντας το ΕΛΚ θεωρώ ότι το επιτελεστά ενέργων της ομάδας εργασίας ε, είναι πολύ ενδιαφέρον έργο, δραστηριοποιήθηκε πολύ ομάδα και θέλω να το υπογραμμίσω και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Όσον αφορά τη στρατηγική, συμπληρώνοντας αυτά που είπατε, τη στρατηγική για την ΤΕΛ, Υπήρξαν δύο εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία, η μία, και στην Πολωνία η άλλη εγκατάσταση. Δεν ξέφυγε κανενός ότι τα προϊόντα που κατασκευόταν στην Ιρλανδία οι υπολογιστές γραφείου ήταν ένα προϊόν που έχανε στην αγορά ενώ όταν άνοιξε το εργοστάσιο της Πολωνίας εκεί ασχολήθηκαν με τους μικροϋπολογιστές και ήταν πιο θετική εξέλιξη αυτού του προϊόντος. Αυτό όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το Ελλανδικό εργοστάσιο. Την άλλη ζητήσαμε ξεχωριστή ψηφοφορία. Το δεύτερο τμήμα όμως απεσύρθη. Όπως επιθυμούσαμε και γι' αυτό ε, συμφωνούμε με το να ψηφίσουμε όλα αυτά μαζί σε ένα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο. Δεν βλέπω. Οπότε προτείνω να ψηφίσουμε το σχέδιο πιστολής για τον πρόεδρο της Επιτροπής Υπολογισμών που ζητά... Α, ο κύριος Καζά θέλει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Φαίνεται ότι συμφωνούμε όσον αφορά την έκθεση. Έχω όμως ένα διαδικαστικό πρόβλημα. Νόμιζα ότι θα ψηφίζαμε στις 5 παρατέταρτο. Ξέρω ότι ο Επίτροπος Αλμούνια είχε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά μας. Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα αυτό σήμερα, αλλά νομίζω ότι όταν έχουμε ένα πρόγραμμα, μια μερίσια διάταξη και έχουμε μια σειρά θεμάτων και συγκεκριμένη ώρα για την ψηφοφορία, πρέπει να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα, διότι πολλοί ευρωβουλευτέ δεν είναι εδώ τώρα γιατί θεωρούσαν ότι θα πρέπει να παραστούν αργότερα. Είναι πολύ κακή συνήθεια στην Οικονομική Νοσηματική Επιτροπή. Θα κάνω ό,τι μπορώ όμως αυτές οι κακές συνήθειε να εξαχθούν στην Επιτροπή Απασχόλησης Λοιπόν, όμως ε, αυτή τη φορά έπρεπε να επιτρέψουμε στον Επίτροπο να παρέμβει αργότερα και εφόσον αφορά ένα κείμενο και είχαμε επίμαχες, επίμαχη ψηφοφορία πολλές τροπολογίες, ε, μπορούσαμε να μετακινηθούμε. Μάλλον θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα όμως συμφώνησαν όλοι χθε, να τα ψηφίσουμε όλα μαζί και δεν νομίζω να υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Δεχόσαστε να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Σας προτείνω να ψηφίσουμε το, την επιστολή για το πρόεδρο της Επιτροπής Υπολογισμών υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται λοιπόν η επιστολή ομόφωνα. Εφόσον συμφωνήσαμε όσον αφορά το σημείο 1, ορίστε, ο κύριος Έλμαρ έχει το λόγο εκτός μικροφώνου και ο Σέλμαρ δεν τον ακούμε. Ενεκρίθη με μία αποχή, όχι ομόφωνα, για την ψηφοφορία, να ψηφοφορία. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ που μας το επισημάνατε. Υπάρχουν άλλες αποχές που μας ξέφυγαν. Ο κύριος Κλάρκ. Όχι αποχή, καταψήφισα. Κυρία Πρόεδρε, ήσασταν πολύ γρήγοροι. Έχουμε μία ψήφο υπέρ, μία κατάλληλη λέει Πρόεδρος και μία αποχή. Το τελικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Στο σημείο 15 προτείνω να εξετάσουμε και να ψηφίσουμε προφορικό, προφορική ερώτηση που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια και που μας επιτρέπει ταυτόχρονα με την εξέταση του αιτήματο κινητοποίησεως του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση στην Ολομέλεια να θέσουμε και το προφορικό ερώτημα άνευ ψηφίσματος και θα μας επιτρέψει γενικότερα να συζητήσουμε το πρόβλημα της μετεγκαταστάσεως των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Ταμείο για την ε, υποστήριξη, για την αντιστάθμιση των φαινομένων των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχουν σχόλια όσον αφορά την προφορική ερώτηση που σας έχει διανεμηθεί. Δεν υπάρχουν σχόλια. Προτείνω να ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε κοινή συζήτηση στην Ολομέλεια πάνω στα δύο αυτά θέματα. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής ερώτησης. Κατά αποχή, ποιος απέχει. Η προφορική ερώτηση εγκρίνεται με μία ψήφο κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξή μας και φτάνουμε στο σημείο 6. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κίνκα Γκόντζ για να αναφερθεί στι τροπολογίε όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη. Κυρία Εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την κινητοποίησή σας. Υπήρξαν ε, πάνω από 100 τροπολογίες. Σχεδόν όλοι ενδιαφερόταν για το θέμα, περίπου 103. Ευχαριστώ για την συνεργασία σας και το επικοδομητικό πνεύμα που επιδείξατε. Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες συναθρίζοντας κάποιες από τις προτάσεις διότι πολλές προτάσεις σχετιζόταν με το ίδιο θέμα και έμοιαζαν πολλοί προτάσεις η μία με την άλλη. Το συζητήσαμε το θέμα με τους κοιόδης ηγητές και όσον αφορά το περιεχόμενο έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε τεράστια προβλήματα Υπάρχει ένα εκρεμές θέμα ακόμα και με τα χαράς να ξανασυναντηθώ με τους σκιώδεις εισηγητές μετά τη συζήτησή μας, τη σημερινή, για να εξετάσουμε την πτυχή της κοινωνικής οικονομίας. Υπάρχουν διάφορα είδη ανησυχιών κατά πόσο τα χρήματα που διατίθενται είναι πολλά ή πολύ λίγα και αυτό συνδέεται με το άνοιγμα του πεδίου που θα καλύπτει τους δικαιούχους ή πόσο θα περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων. Αυτό που το συζητήσουμε περαιτέρω. Υπάρχουν δύο άλλα εκρεμή ζητήματα. Το ένα αφορά τις ε, εθνικές μονάδες και έχουμε τροπολογία για μηχανισμό της αξιολογήσεως των δράσεων μικροοικονομικής μικροχρηματοδοτήσεων σε εθνικό επίπεδο. Υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν κάποιες αντιστάσεις από κάποια κράτη-μέλη. Έλεγαν ότι δεν πρέπει να συμπεριλάβουμε κινήσεις σε αυτό το επίπεδο, μην αυξήσουμε τη γραφειοκρατία. Να επιτραπεί κάτι τέτοιο, εθνική ρύθμιση για κάποιες χώρες, αλλά να μην είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να μην ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο. Το βασικό πρόβλημα είναι οι πόροι. Ίσως ε, γνωρίζετε, συζητούμε κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιούμε νέους πόρους ή πόρους του Progress ή εν μέρη πόρους του Progress για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επανειλημμένα επιχειρηματολόγησα λέγοντας ότι όλη η φιλοσοφία του προγράμματος διαφέρει από τη φιλοσοφία του Progress μπορεί να προσελκύσει πόρους από τράπεζες από την αγορά Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε νέους πόρους που απορρέουν από αυτή τη φιλοσοφία. Το Κοινοβούλιο από την άλλη ψήφισε να αυξηθούν τα κονδύλια για το Progress. Και τώρα να πάρουμε πόρους από το Progress δεν θα ήταν κάτι αποδεκτό το Κοινοβούλιο. Και το Progress και το νέος μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων εστιάζονται στα, στους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα. Εν μέσω κρίσεως δεν θα πρέπει να αφαιρέσουμε χρήματα που έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Ε, θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότηση. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις του ΕΛΚ να αφαιρεθούν κάποια χρήματα από το Progress, αλλά η Οικονομική Επιτροπή υποστηρίζει τη δική μας προσέγγιση. Και από ό,τι γνωρίζω, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και ο πρόεδρος Επιτροπής αυτής υποστηρίζει τη θέση μας. Δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τα νέα προγράμματα, λένε. Θα ήθελα να ξέρω εσείς τι πιστεύετε. Γιατί είναι η μεγάλη εκκρεμότητα για μας. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν και ποια είναι η άποψή σας για τις τροπολογίες, τις άλλες. Προσπάθησα όσο μπορούσα να πετύχω συμβιβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας και για τη συνεργασία σας. Πολύ ωραία. Ποιος θέλει το λόγο? Ο κύριος Σέρκας. Κύριε Σέρκας, πριν σας δώσω το λόγο, συγχαρητήρια για τα χθεσινά MEP Awards για το βραβείο. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και σε εσά για την υποψηφιότητά σας. Και είμαι βέβαιος ότι του χρόνου στη δική σας γιορτή θα πάρουμε μέρος. Θα ήθελα να υποστηρίξω την εισηγήτριά μας. Συμφωνώ μαζί της και θα ήθελα να υπενθυμίσω κυρίως τους νέους ευρωβουλευτές ότι στη συζήτηση αυτή προσπίσουμε μια ιστορική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επετέχθη με συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων. Και ήταν επίπονη διαδικασία αυτή η χρηματοδότηση του μηχανισμού. Και προσπαθούν τώρα από την Κερκόπορτα να ακυρώσουν μια τέτοια απόφαση. Δίνουμε μάχη λοιπόν για να αυξήσουμε τον προπολογισμό του Progress και δεν μπορούμε με ένα τέτοιο πολιτικογραφιοκρατικό ελιγμό να υπονομεύσουμε τις προτάσεις μας. Η εισηγήτρια επίσης έχει δίκιο που υποστηρίζει ότι μεσούς της κρίσης πώς είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε ότι η αλληλεγγύη προς τους πλέον άπορους θα πρέπει να προκύψει από τους άλλους ε, δικαιούχους της ε, κοινωνικής στήριξης. Θα πρέπει ε, από αλλού να προκύψει τα κονδύλια και όχι εις βάρος άλλων δικαιούχων. Δεν μπορούμε να ζητούμε χρήματα από ένα φτωχό για να βοηθήσουμε άλλον. Θα πρέπει να γίνει ένας καλός συντονισμός των πόρων, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει αυτό εις βάρος άλλων προγραμμάτων αλληλεγγύης για να χρηματοδοτηθεί αυτός ο μηχανισμός της αλληλεγγύης. Υπάρχει μια τροπολογία του ΕΛΚ που είναι αρκετά λογική και που λέει ότι ας γίνει ένας επιμερισμός, ας γίνει μια κατανομή. Ούτε όλο το progress, αλλά ούτε να, μην δεχτούμε ούτε ένα μικρό του progress. Θα δούμε πώς ε, θα χρηματοδοτηθεί, θα χρηματοδοτηθεί αυτός ο νέος μηχανισμός. Ίσως ε, με ένα συνδυασμένο σύστημα, ένα μεικτό σύστημα. αλλά δεν θα πρέπει να ανοίξουμε όλα μας τα χαρτιά. Θα ήθελα να πω στα μέλη του ΕΛΚ ότι παρόλο που πιστεύουν ότι μπορεί αυτή να είναι η τελική λύση, να μην υπονομεύσουν τώρα τη διαπραγματευτική μας ισχύ. Θα μπορούσαμε τώρα να υιοθετήσουμε σε διαπραγματευτική θέση ότι τίποτα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα και αργότερα σε μεταγενέστερη φάση της διαπραγμάτευσης ίσως χρειαστεί να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκε το ΕΛΚ, η κυρία Μο... και μετά η κυρία Σρέτερ. Σιρέτερ. η κυρία Σρέτερ και μετά η κυρια σιρετερ και Μωρά, όπως προτιμάτε. Äh, ναι, ήθελα πάνω να ξεκαθαρίσω το εξή, ότι πήραμε μία απόφαση στην Ολομέλεια κατά την πρώτη ανάγνωση του προπολογισμού, όπου η θέση του Κοινοβουλίου ξεκαθάρισε πλέον. Δεν έχει λοιπόν νόημα να προσπαθήσουμε εδώ στην Επιτροπή να αλλάξουμε την απόφαση αυτή που πήρε η Ολομέλεια, γιατί αποδυναμώνουμε έτσι την θέση των διαπραγματευτών σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό ανεξάρτητα από τα μεμονωμένα προβλήματα. Το γεγονός, το θέμα του πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα, θα το εξετάσουμε αργότερα και θα το αποφασίσουμε αργότερα. Δώσαμε ως συντονιστές ε, εντολή για ενέργεια έρευνας για να δούμε τον αντίκτυπο των μικροχρηματοδοτήσεων και έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε τα μέσα αυτά. Καταρχάς, το θέμα είναι η γραμμή του προϋπολογισμού, αυτά που δημιουργήσαμε, αυτά που ψηφίστηκαν στην Ολομέλεια, να έχουν νομική βάση. Γι' αυτό λοιπόν η ψηφοφορία αυτή θα πρέπει να περιοριστεί στο περιεχόμενο της νομικής βάσης, τους όρους για την δαπάνη των κονδυλίων. Όχι να ξαναθέσουμε εκ νέου αυτό το βασικό θέμα, το βασικό ερώτημα αν θέλετε. Ε, Η κυρία Μοάχαν και μετά ο κύριος Σέλμαρ. Άκουσα με προσοχή την εισηγητριά μας και τις παρατηρήσεις του Αλεχάνδρου Σέρκας. Καταρχήν, το γεγονός ότι τροποποιήσαμε πολύ γρήγορα στην αρχή της συνεδρίασης τη σειρά των σημείων συζήτηση ημερήσιας διάταξης ε, Μα στέρισε από την αρχή την παρουσία του σκιώδου μας συγητού. Που στο μεταξύ έφτασε όμως, καλό θα ήταν λοιπόν να τον ακούσουμε. Είναι αναφίβολο πάντως ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι σκόπιμο να αναπτύξουμε αυτό το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων. Όλοι θέλουμε αυτό το μηχανισμό και ο Αλεχάνδρος Σέρκας είπε ότι με αυτό το στόχο συμπαρατάχθηκαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια υπάρχει ίσως κάποια διάσταση απόψεων ως προς τους τρόπους υλοποίηση αυτού του στόχου, αν και ως προς το στόχο συμφωνούμε. Επί της ουσίας λοιπόν είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι χρειαζόμαστε μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων, κυρίως για να βοηθήσουμε τους πλέον άπορους σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Αλλά όταν μιλούμε για νέα κονδύλια, για φρέσκο χρήμα, προβληματίζομαι. Γιατί ακριβώς επειδή διανύουμε μια κρίση, έχουμε ένα πολύ λιτό προϋπολογισμό. Και γι' αυτό οι θέσεις μας ως προς τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι πολύ υπεύθυνοι. Και η αλληλεγγύη που θέλουμε να δείξουμε δεν θα πρέπει επουδενή να μας οδηγήσει σε μη βιώσιμες δημοσιονομικές λύσεις. Θέλουμε λύσεις που και από οικονομική και άποψη δημοσιονομική θα είναι εφικτές και βιώσιμες δεδομένου του σχετικά περιορισμένου μας προϋπολογισμού. Και με αυτή τη λογική θα ψηφίσουμε όλα, Γιατί δεν θέλουμε να λάβουμε θέσεις που θα έρχονται σε αντίθεση με την ευθύνη ενός ε, Ευρωβουλευτή να ψηφίζει έναν ε, εφικτό προϋπολογισμό. Εδώ βλέπω τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης είναι ακόμη πιο αυστηρά και απαιτητικά από τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση προδιαγράφεται και θα συνεχιστεί και με τον Επίτροπο Αλμούνια. Ο κύριο Έλμαρ και μετά η κυρία Χάρκιν. Um, κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την προηγούμενη ομιλήτρια και την κατεύθυνση που ακολουθεί. Το έχω σχολιάσει πολλέ φορέ και θα το επαναλάβω ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε όλο τον κόσμο οι εθνικέ κυβερνήσει αντιδρούν στην οικονομική κρίση προσπαθώντας να ελέγξουν και να μειώσουν τις δαπάνες τους. Και νομίζω ότι ο κόσμος όπου μας εξέλεξε το θεωρεί ότι περίεργο. Γιατί οι κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο προσπαθούν να περιορίσουν τις δαπάνες και εμείς ε, αντιδρούμε στην κρίση απαιτώντας πιο πολλές δαπάνες. Θεωρώ ότι και οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί ε, αντιτίθενται στην διάθεση περαιτέρων πόρων. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεταφορά 50 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Progress στο, στις ε, μικροχρηματοδοτήσεις και προετοιμάσαμε την υποστήριξή μας χωρίς μεγάλο ενθουσιασμό για το πρόγραμμα αυτό. Ωστόσο, δεν θα υποστηρίξουμε άλλες δαπάνες. Ανησυχούμε, στόσο λίγο για τις συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες δεν προετοιμάστηκαν μάλλον δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε όσο έχουν, ιδιαίτερα επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπός είναι να υποστηριχθούν μικρά προγράμματα, τα οποία έχουν κάποια προπτική επιτυχίας. Αν με τις συμβαστικές τροπολογίες αυτές αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και αν επικεντρωθούμε όμως στα άτομα αυτά που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και αποκλείονται από το συμβατικό χρηματοπιστωτικό πρόγραμμα, ουσιαστικά είναι σαν να υποστηρίζουμε προγράμματα με λιγότερε πιθανότητε επιτυχία. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι ανεπιθύμετο. Δεν θα υποστηρίξουμε λοιπόν τι τροπολογίε αυτέ. Ευχαριστώ. Κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. καταρχά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία μας καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και πραγματικά θα ήμουν υπέρ των συμβαστικών τροπολογιών. Νομίζω ότι θέτει κάτι το πολύ σημαντικό όταν λέει ότι μιλάμε για ανακυκλούμενους πόρους. Δεν τα επενδύουμε και δεν θα τα χάσουμε και νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε πιο πολλούς πόρους και τέτοια χρήματα. Υποστηρίζω την εισηγήτρια λοιπόν επί της βάσεως αυτής. Έχω ωστόσο δύο-τρία ερωτηματικά. Μία ερώτηση είναι η εξή. Είναι πιθανό να καθυστερήσει έτσι η εφαρμογή του Ταμείου. Μπορούμε να το πούμε αυτό σήμερα ή είναι κάτι το οποίο θα φανεί στο μέλλον. Και κάτι άλλο το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμα. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα επιτροπολογίας και τροποποίησης ε, της απόφασης από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν ε, ξέρω αν θα το συζητήσουμε εδώ και φυσικά αυτή η απάντηση θα πρέπει να ληφθεί πρώτα από το Κοινοβούλιο, δεν μπορώ να τη συζητήσω εγώ. Τελευταίο σχόλιο, μάλλον δύο τελευταία σχόλια. Καταρχάς, και δεν έχει ξαναναφερθεί και αυτό, η επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας μπορεί να επηρεάσει το θέμα αυτό. Και τέλος, αυτά που είπε ο τελευταίος ομιλητής ε, για τις κυβερνήσεις που προσπαθούν να ελέγξουν και να περιορίσουν τα έξοδά τους. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για μια επένδυση, μια επένδυση σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν άλλη πρόσβαση σε πίστοση. Δεν μιλάμε μόνο για την επιτυχία των επιχειρήσεων, δεν είναι μόνο αυτό το πιο σημαντικό. Μιλάμε και για θέματα κοινωνικής συμμετοχής. Αυτό έχει πολύ ευρύτερο αντίκτυπο και ως Κοινοβούλιο θέλουμε να διασφαλίσουμε ε, άτομα ή ε, οργανώσεις που δεν έχουν ε, άλλη πρόσβαση σε πιστώσεις γιατί δεν τους δανείζουν οι τράπεζες. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα αυτά θα έχουν πρόσβαση στην πίστοση, σε πιστώσεις. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν φυσικά και κάποιοι κάποιες ε, προδιαγραφές. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο φατική η στάση μας από ό,τι αυτή που περιγράψατε. Ευχαριστώ κυρία Σιλβάνα Αράπτη και μετά κύριο Σούγκερα Κυρία Αράπτη. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ε, θέλω να δώσω πρώτα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια την Κίνκα για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Δεύτερον, θέλω να δηλώσω ότι βρίσκομαι σε ευθεία γραμμή με το σκεπτικό που ανέπτυξε ο κύριος Σέρκας και τρίτον, θέλω να επισημάνω ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε μία απόφαση την οποία παίρνουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι το πρόσωπο της κοινωνικής Ευρώπης, το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης κοντεύει να εξαμφανιστεί, νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το να πάρουμε χρήματα από τους λιγότερο φτωχούς για να τα δώσουμε στους περισσότερο φτωχούς δεν νομίζω ότι μας οδηγεί στο ποθητό αποτέλεσμα νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στους ανθρώπους αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και που δίνοντα τους χρήματα αυτά θα επανέλθουν σε εμά, θα επανέλθουν στο κοινωνικό σύνολο μέσα από μια άλλη διάσταση. Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και κλείνοντα επισημαίνω ότι για μένα δεν θα πρέπει τα χρήματα να προέλθουν από το Progress. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να υποστηρίξω και εγώ τη συνετή οικονομική προσέγγιση. Ναι, καλή αυτή η μικροχρωματοδότηση αλλά νέα χρήματα, φρέσκα χρήματα, νέες πιστώσεις είναι αυτό που ζητάμε. Αλλά αυτό ίσως να πιέσει περισσότερο τα περιθώρια του προπολογισμού και πολλά πιλωτικά προγράμματα θα κινδυνεύσουν τι ούτω τρόπος. Νέα χρήματα ίσως να σημάνει μη πιλωτικά προγράμματα. Αν ευπροηγουμένου πίεση ασκείται στα αποθεματικά του προπολογισμού, όπως χρήματα που χρειάζονται για να σταματήσει η λειτουργία του Κοσλοντούι. Χρειάζεται 300 εκατομμύρια ευρώ αυτή η δουλειά. Από το 2010 μέχρι το 2013 για να κλείσει το Κοσλοντούι. 75 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο θα βγαίνουν από το αποθεματικό και θα μείνουν περίπου 37 εκατομμύρια θα μένουν στο αποθεματικό. Το να φερούμε χρήματα από το αποθεματικό λόγω αυτό του περιβάλλοντος τεραστίων πιέσεων που ασκούνται στα αποθεματικά νομίζω ότι δεν είναι η πιο συνετή προσέγγιση. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Εγώ ε, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την ομάδα που δεν ανήκω και κυρίως εντό του ΕΛΚ, τι διευθετήσεις γίνονται. Εκπλήσω όμως από τον τόνο της συζητήσεως που διαμορφώνεται στη δική μας Επιτροπή, διότι στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή η ομάδα του ΕΛΚ ψήφισε στο πνεύμα αυτό της εισηγήτριάς μας. Στην Επιτροπή Προπολογισμών μου λένε ότι το ΕΛΚ ετοιμάζεται να υποστηρίξει την ίδια στατηγική. Επί της ουσίας, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στην επιχειρηματολογία. Όσον αφορά την χρήση χρημάτων που βγαίνουν από το αποθεματικό, είναι πραγματικά φρέσκα χρήματα, νέα χρήματα που θα επηρεάσουν κάπως τη διαχείριση των χρεών των κρατών μελών ή το έλλειμμα του προπολογισμού. Μπορούμε να αρχίσουμε τώρα θεωρητική συζήτηση. Αλλά εδώ δεν έχουμε φρέσκα χρήματα. Χρησιμοποιούμε τα περιθώρια, τα αποθεματικό. Όσον αφορά την ουσία, βλέποντας τα αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης, όταν συζητήσαμε τον προπολογισμό στο Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο έναντι της κρίσεως που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο καθόρισε τις προτεραιότητες. Τη χρηματοδότηση του δεύτερου τμήματος του σχεδίου ανάκαμψης, τη διαχείριση της κρίσεως του τομέα του γάλακτος και αυτό το πρόγραμμα για τη μικρή χρηματοδότηση. Είναι ένα πρόγραμμα που ψηφίστηκε σαν μία από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις στη συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό. Και εγώ πρέπει να πω ότι θα έβρισκα άκρος παράδοξο το ότι η Επιτροπή ασχολείται, που ασχολείται επί της ουσίας με αυτό το θέμα είναι κατά για θέματα, για λόγους του υπολογισμού. χρησιμοποιώντας επιχειρήματα άλλης επιτροπής που εκείνη η άλλη επιτροπή είχε υποστηρίξει τα εν λόγω προγράμματα, το εν λόγω πρόγραμμα. Και έχουμε και τρίτο θέμα, τρίτο επιχείρημα. Μέσα σε μια κρίση Υπάρχουν δύο στάσεις. Να μπει κανείς με σπίτι του, να κλείσει την πόρτα του, να μην τρώει και να περιμένει να περάσει η κρίση. Αυτή είναι η μία στάση. Η άλλη στάση είναι να ανοίξει την πόρτα και να προσπαθήσει να βρει άλλου, να δει αν μπορεί να κάνει κάτι και αν μπορεί να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει. Και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα της μικροχρηματοδότησης αντιστοιχεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική. Δεν έχουμε τόσα παρόμοια εργαλεία στη διαθέσή μας για να προχωρήσουμε αύριο. Αυτό το πρόγραμμα είναι προς τιμήν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι υπέρ των πλέον ευαλώτων συμπολιτών μας. Και φανταστείτε ότι επειδή θα χρηματοδοτήσουμε αυτό, να υπαναχωρήσουμε από ένα πρόγραμμα που, για το οποίο πολέμησε στεναρά το κοινοβούλιο αυτό και η επιτροπή αυτή στα πλαίσια του Progress. Αν το κάνουμε αυτό θα είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Και αν αυτό το κοινοβούλιο μετά από αυτές τις εκλογές στο κλίμα που βρισκόμαστε στείλει ένα μήνυμα από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που αρνείται να εξετάσει σοβαρά την εφαρμογή αυτού του εργαλείου που πωλείται σαν, ένα, σαν μια απάντηση στην κρίση, αν γίνει αυτό, νομίζω ότι θα είναι πολύ εσφαλμένο και ο καθένας μπορεί να κρίνει στη συνείδησή του και στην ψυχή του τη θέση του και νομίζω ότι η νύχτα θα είναι καλός σύμβουλος. Το ξανασκεφτείτε. Δεν έχω άλλους ε, ομιλητές στον κατάλογο μου. Η κυρία να έχει το λόγο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια σχολιάζοντας ε, τη δική σας σύνοψη. Αυτό που είπα για το ΕΛΚ και αυτό που είπε η συγκεκριά μας δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία. Ως προς την ουσία, ως ως προς τον πολιτικό στόχο και το στρατηγικό στόχο των μικροχρηματοδοτήσεων συμφωνούμε. Υπερψηφίσαμε αυτή την πρόταση και την στηρίζουμε. Και είμαστε υπέρ και δίνουμε μάχη χρόνια ολόκληρα στην Επιτροπή αυτή υπέρ της ε, ένταξης, της κοινωνικής ένταξης, ε, της επαγγελματικής ένταξης και ο, μικροχρημα... μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων είναι ένα από τα μέσα ένταξης και ανέκαθεν ε, είχε τύχει της υποστήριξής μας. Αλλά ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Γιατί εσείς αναφερθήκατε στο στόχο και εγώ αναφέρθηκα στα μέσα για την υλοποίηση του στόχου. Εκεί είναι που διαφέρουμε. Οι στόχοι μας είναι κοινοί. Αλλά ο τρόπος υλοποίησής τους είναι διαφορετικός. Αλλά μπορείτε να μας έχετε εμπιστοσύνη κυρία Πρόεδρε γιατί και εμείς θα επιδιώξουμε τον κοινό μας στόχο. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Η για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και για την πολύ ζωηρή συζήτηση που έγινε για το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων. Μόλις το πρωί είχαμε συζήτηση με την ε, Επιτροπή για την κρίση και εκεί αναφέρθηκε κάτι πολύ σημαντικό Είπαμε ότι θέλουμε περισσότερο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη και αυτό προσπαθούμε να ενισχύσουμε. Να βοηθήσουμε εκείνους που δεν έχουν ούτε τις δεξιότητες, ούτε τις γνώσεις, να στραφούν στην αγορά και να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες, κάποια προσόντα και να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις, μικροεπιχειρήσεις που θα είναι και βιώσιμες. Και αυτό αναφέρθηκε και για το τρόπο παροχής συμβουλών, το mentoring, που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, θέλουμε να αποφύγουμε χρονοτριβές στην εφαρμογή του προγράμματος. Ευελπιστώ ότι ο τριμερής διάλογος θα αρχίσει το αργότερο 16 Νοεμβρίου. Και όπως άκουσα από προηγούμενες συζητήσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, υπάρχει ε, μια διαλλακτικότητα προς τα δικά μας επιχειρήματα και το περιθώριο ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων. Καλό θα ήταν να αναμίξουμε και μη συμβατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να χρηματοδοτήσουμε και από εκεί το μηχανισμό. και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ μικρό τμήμα των κονδυλίων του Progress για αυτό το capacity building, για την ε, ενίσχυση του δυναμικού. Αλλά όχι όλο το πρόγραμμα, όχι όλος ο προϋπολογισμός να, προέλθει, να προέλθει από το Progress. Η κυρία Μαρία Χάρκιν μίλησε για χρήματα που επιστρέφουν ουσιαστικά. Είναι κονδύλια που θα επανέλθουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και θα πρέπει να βρεθούν και πόροι για το πακέτο ανάκαμψης που είναι 2,5 δισεκατομμύρια και όχι 37,5 εκατομμύρια. Οπότε από αυτήν την άποψη ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων δεν είναι και τεράστιο κονδύλιο και μπορούμε πιστεύω να το χρηματοδοτήσουμε από το περιθώριο. Ελπίζω να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος το συντομότερο δυνατό ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα και αυτό τάχιστα. Περιμένουμε και την έκθεση της Μαρίας Χάρκιν που θα συζητήσουμε σε λίγο και θα πρέπει να περιμένουμε και αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να προσθέσω ότι το ΕΛΚ 100% υποστηρίζει το πρόγραμμα για τις μικραχρωματοδοτήσεις, αλλά θέλουμε να βρούμε και έναν αρθολογικό τρόπο να χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι δεν είναι θέμα του αν θα γίνει το πρόγραμμα αυτό, το θέμα είναι το πώς θα εκτελεστεί. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αυτό για τη θέση μας. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το σημείο 6 για να ικανοποιήσουμε και τον κύριο Κάζα θα ψηφίσουμε αύριο για το θέμα αυτό από τις 9 και μετά όπως είχαμε συμφωνήσει αρχικά θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε αύριο οπότε η έκθεση αυτή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Πέραμε τώρα στο σημείο 8. Εξέταση της της κυρίας Μάριαν Χάρκιν με θέμα το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, που θα είναι το 2011. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θα ήθελα να την ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά συμφώνησε με αυτούς τους εξαιρετικά σκληρούς όρους ε, του χρονοδιαγράμματος. Γιατί ενώ από την αρχή της θητείας το χρονοδιάγραμμα ήταν κάπως αβέβαιο, τον τελευταίο καιρό επιταχύνθηκε κάτι που πίεσε αφόρητα τη συντάκτρια της γνωμοδότης προκειμένου να εκπονήσει έγκαιρα τη γνωμοδότησή της για να την διαβιβάσει την αρμόδια καθήλη επιτροπή. Αλλά παρόλα αυτά τα κατάφερε η Μαρία Χάρκιν και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στο χρονοδιάγραμμα και για να κατατοπίσω και τα μέλη να σας πω ότι βρισκόμαστε σε φάση διαβούλευσης και ο λόγος που αποφασίσαμε να επιταχύνουμε την διαδικασία και να συνεργαστούμε με τον εισηγητή τον κύριο Σκούρια είναι ότι η Σιωτική Προεδρία εγγυήθηκε ότι θα υπήρχαν πραγματικές διαβουλεύσεις, ότι θα λάμβαναν υπόψη δηλαδή τις θέσεις του Κοινοβουλίου, γιατί φυσικά μετά την Λισαβόνα, μετά τη Λισαβόνα θα ακολουθηθεί η διαδικασία της συνένεσης, δηλαδή το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πει ναι ή όχι, χωρίς να επηρεάσει τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό λοιπόν επιταχύναμε τη διαδικασία, αλλά αρχικά νομίζω υποτίθεται ότι θα πήγαινε στην Ολομέλεια τον Δεκέμβριο. Ε, από όσο καταλαβαίνω, εκτός και αν καταφέρουμε να το κάνουμε τον Νοέμβριο, θα ε, ουσιαστικά υπαχθεί στην συνθήκη της Λισαβόνας, θα αλλάξει η νομική βάση. Αλλά αυτό να το αφήσω και στους ειδικού. Όπως σας είπα, ο κύριος Κούρια μας ανακοίνωσε ότι ήταν διατεθειμένος να συμμετάσχουν στις ισχυώδεις εισηγητές ε, στις ε, συνεδριάσεις με τους ειδική προεδρία. Ε, επικοινωνήσαμε με το γραφείο του, δεν πήραμε απάντηση και αποφάσισα να μην το ξαναζητήσω, να μην το ξαναθέσω αυτό το θέμα μέχρι να το συζητήσουμε και στην Επιτροπή. Ελπίζω ωστόσο να ισχύσει αυτό γιατί θα είναι πραγματικά ωφέλιο, ωφέλιμο. Δύο γενικά σχόλια για τις τροπολογίες και του κυρίου Σκούρια. Κάποιες είναι σημαντικές για την Επιτροπή μας. Για δύο συγκεκριμένες τροπολογίες, την 4 και την 11. Αλλάζει εκεί ο εισηγητή τη φράση professional skills, επαγγελματικές ικανότητες. Το κάνει οι κοινωνικές ικανότητες και αντί για οικονομική ε, συνοχή μιλάει για κοινωνική συνοχή. Και αυτό το αλλάζει και μου φαίνεται ότι αλλάζει, αν θέλετε, την κατεύθυνση, γιατί θεωρώ ότι και η οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτελούν τμήμα της έκθεσης. Και επίσης, αυτό το λέω ως γενικό σχόλιο. Πέραν αυτών, έγινε μια συνάντηση με τους περισσότερους κοιόδης σήμερα το πρωί ήταν πραγματικά εξαιρετική η συνάντηση αυτή και καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για όλα σχεδόν τα θέματα για τις τροπολογίες και ελπίζω όταν λάβουμε τις τροπολογίες να τις ε, κοιτάξουμε σήμερα το απόγευμα. Ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχουν ε, ιδιαίτερα πολλά έκρεμη ζητήματα. Να κάνω κάποια σχόλια για τις δικές μου τροπολογίες και θα είμαι σύντομη. Η πρώτη τροπολογία προτάθηκε για να ενισχυθεί η νομική βάση πολύ απλά. Άλλε τροπολογίε που θεωρώ ότι είναι σημαντικέ. είναι να συμπεριληφθεί η διάσταση της συμμετοχικής δημοκρατίας που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τον εθελοντισμό. Επίση, η συμπερίληψη του εθελοντισμού μεταξύ των γενεών και επίσης να διασφαλιστεί ο εθελοντισμός προωθεί τον ε, κοινωνικό την κοινωνική συμμετοχή, την καταπολέμηση του ρατσισμού και επίσης τον διαεθνικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Ένα άλλο σχόλιο είναι το εξής. Υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες και ευκαιρίες συνέργειας με διάφορα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα φέτος, αλλά και με τους ε, Ολυμπιακούς, τους ειδικούς Ολυμπιακούς του 2010 στην Αθήνα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πραγματικά πολλές ευκαιρίες για να τονώσουμε και να υπογραμμίσουμε τη σημασία του εθελοντισμού και για να αναγνωριστεί η αξία του. Ένα άλλο θέμα το οποίο ανέφερα ήταν η οικονομική αξία του εθελοντισμού. 31 χώρες έξι εξ αυτών είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούν το εγχειρίδιο του ΟΗΕ που προσμετρά την συμμετοχή, τη συμβολή του αθλητισμού, όπως το Βέλγιο και η Ουγγαρία. Αυτό τι καταδεικνύει ότι ανέρχονται το κέρδος σε 5 8% Άρα, οι πιο πολλοί συνειδητοποιούν την κοινωνική διάσταση του εθελοντισμού, αλλά είναι σημαντική και η οικονομική διάσταση και αυτή αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα ε, της ε, συνολικής εξίσωσης και έχουν συμφωνηθεί και με τον Τζον Χόπκινς και με την, τον ΟΙΕ να εισαχθεί αυτή η μέτρηση του εθελοντισμού, η συμβόλη του εθελοντισμού μέσω των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι έχει, σημαντηθεί, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο. Γιατί για πολλού ξέρετε, αν δεν μπορεί κανεί να δώσει έναν αριθμό, ε, δεν μετράει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, θεωρώ, αυτό μια άλλη πτυχή του εθελοντισμού. Δύο άλλα στοιχεία. Ζήτησα να αυξηθεί ο προπολογισμό από 6 σε 12 εκατομμύρια, κοιτώντα κάποιε άλλε χρονιές, μάλλον ευρωπαϊκέ ε, χρονιές, ε, αφιερωμένες θέματα, θα δείτε ότι είναι πολύ πιο, πολύ πιο μεγάλη, ο μεγάλος ο προπολογισμός. Επίσης, απέσυρα τις τροπολογίες για να καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 80%. Ε, εγώ είχα βάλει 75%, αλλά τέλος πάντων μετά από τη συζήτηση με άλλους ε, σκιώδεις συνειδητοποιήσαμε ότι το επίπεδο της χρηματοδότησης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε κάποιες χώρες και δεν το επιτιμούσαμε φυσικά αυτό, άρα δεχτήκαμε το 80%. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Συγκήτρια. Η κυρία Γιούτα Στάινρουκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για την ε, πολύ καλή και ισοσκελισμένη έκθεση και για την συνεργασία μας που ήταν πολύ επικοδομητική. Ήταν πραγματικά η πρώτη τέτοια ευχάριστη συνάντηση που είχαμε. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Μία κοινή τροπολογία με τους πρασίνους για την διασφάλιση σε περίπτωση ατυχημάτων. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ε, σε περίπτωση ατυχημάτων θελοντών να είναι ασφαλισμένοι οι θελοντές και οι ίδιοι και για την αστική τους ευθύνη. Επίσης, ό,τι αφορά τις ε, συνταξιωτικέ απαιτήσεις, Η εμπειρία μας από τη Γερμανία καταδεικνύει ότι ε, η εθελοντική εργασία ε, είναι δυνατόν να σημαίνει και συνταξιωτικά δικαιώματα. Και αυτό το παράδειγμα θα θέλαμε να το μεταδώσουμε και σε άλλες χώρες ως ένα τμήμα των βέλτιστων πρακτικών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Καρίν Μπαντελή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σαν συγγήτρια της ε, Επιτροπής Περιφερικής Αναπτύξεως πρέπει να πω ότι ψηφίσαμε την έκθεση σήμερα το πρωί και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Άρκιν για τη δουλειά που έκανε και για τη συνεργασία της κυρίως στο πλαίσιο αυτό που δεν πήγαν κάτα πράγματα για τον εθελοντισμό. Μας λέγανε ότι πρέπει να περιμένουμε τη Λισαβόνα και μετά έπρεπε να ασκηθεί κάποια πίεση από τη Σουηδική Προεδρία που ήθελε να συμπεριλάβει το θέμα στο έργο της και λοιπά. Μελέτησα προσεκτικά τις τροπολογίες και πιστεύω πραγματικά ότι αυτές που υπέβαλε η κυρία Χάρκιν εμπλουτίζουν πράγματι το κείμενο και από πλευρά αύξηση των κονδυλίων και προστασία των εθελοντών και την προστασία της αξίας του εθελοντισμού. Αλλά ήθελα να διευκρινίσω ότι καταθέσαμε και κάποιες τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα μια τροπολογία η οποία θα τονίζει τα κριτήρια που τίθενται από τον ΙΕ και το Εθνές Γραφείο Εργασίας και που διευκρινίζει που, διευκρινίζει τι είναι ο εθελοντισμός. Το έτος εθελοντισμού θα πρέπει να ενθαρρύνει κάθε χώρα να δημιουργεί πραγματικά ένα καθεστώς για τους ε, εθελοντές. Αλλά να πρέπει να υπάρχουν να προβλέπονται και συνθήκες εργασίας. Το δεύτερον, δεν πρέπει ο εθελοντισμός να αντικαθιστά μία μισθωτή ε, δραστηριότητα διευκρινίζω, οι κρατικές αρχές δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την εθελοντική εργασία για να αντικαθιστούν με μικρότερο κόστος λειτουργίες που ε, αφορούν τις δικές τους υπηρεσίες και την δίκηση γενικά. Ε, μετά, όπως είπε η κυρία Χάρκιν, υποβάλλουμε τροπολογία για να πούμε ότι το έτος εθελοντισμού είναι ένα έτος αλληλεγγύης, ένα έτος συνεργασίας, μια χρονιά καταπολέμησης κάθε διάκρισης λοιπόν και πρέπει να είναι προσβάσιμο το καθεστώς αυτό σε όλους τους, που, ξένους που διαμένουν σε κάθε κράτος μέλος. Μετά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί αυτό το έτος, μπορούμε να το κάνουμε αν αγγιηθούμε αποτελεσματική προστασία υγείας και ασφαλείας τους εθελοντές. Εξηγούμε σήμερα πολλοί εθελοντές πηγαίνουν σε εργοτάξια, καμιά φορά σε εργοτάξια που έχουν αμύαντο και δεν προστατεύονται ή οι εθελοντές πυροσβέστες. Θα πρέπει να προβλέπετε μια προστασία της υγείας τους και της ασφαλείας τους. Και τέλος, το έτος του εθελοντισμού, όπως υπενθυμίζει και μια έννοια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι η πρόθεση της ειρήνης. Αυτή η χρονιά θα πρέπει να δείχνει ότι ο εθελοντισμός επιτρέπει την πρόθεση της ειρήνης, αλλά όχι μόνο αυτό, αφορά ανταλλαγή λαών, συνεργασία βορρά-νότου, και πρέπει να επιθυμήσουμε την αλληλέγγυα και κοινωνική οικονομία. Πρέπει να προβάλλεται αυτή η οικονομία. Ευχαριστώ. Σότσο Βάσκορ. Σας ευχαριστώ. Είμαι ο εισηγητής εκ μέρους του ΕΛΚ και συμφωνήσαμε για όλα τα στοιχεία της γνωμοδότησης. Έχουμε υποβάλει και κάποιες προτάσεις τροπολογίες. Και μάλιστα είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του θελοντισμού και της έμης της δραστηριότητας. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο ενιών. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις νέες δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί η χρηματοδότηση δημιουργεί προβλήματα. Και συμφωνήσαμε με το διπλασιασμό του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Γιατί σε αυτές τις νέες δημοκρατίες η κοινωνία των πολιτών και εθελοντισμός είναι ε, νέες εμπειρίες ε, αρκετά ευάλωτες και καλό θα ήταν ο εθελοντισμός να μην περιοριστεί μόνο στο 2011 αλλά να γίνει μια μόνιμη πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει άλλος κανείς το λόγο παρακαλώ. Ουδής δεν υπάρχει και εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Συγγήτρια, έχετε το λόγο αν το επιθυμείτε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες οι περισσότεροι, συμφωνούμε σε πολλά σημεία. Αναφέρθηκε το θέμα της ασφάλειας για ατυχήματα, ασφάλειας ε, υγείας και ζωής. Επίσης το θέμα των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Θα φροντίσουμε να βρούμε μια τροπολογία και γι' αυτό. Επίσης, ε, διαφορά μεταξύ του Βολονταριά και του Μπενεβόλα αυτό υπάρχει σε ορισμένες χώρες, ε, γιατί στις περισσότερες υπάρχει ένα ενιαίος εθελοντισμός. Θα μπορούσαμε να βρούμε πάντως ένα πλαίσιο που να ικανοποιεί τις χώρες που έχουν αυτή τη διάκριση. Επίσης, να μην αντικαταστήσουμε την έμιστη δραστηριότητα με τον εθελοντισμό. Και εθελοντικές δραστηριότητες ε, δεν θα πρέπει, και που λέμε δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν έμιστες, να πούμε ε, δεν πρέπει ε, δεν, γίνεται, δεν, δίν, δεν δίνονται να αντικαθιστούν έμιστε. Στο σημείο 11 μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, το should από το must. Σας ευχαριστώ. Κύριε Συγκήτρια, έρχεται μέχρι το τέλος της ημέρας για να εκπονήσετε και τις τελευταίες συμβαστικές προτάσεις. Η κυρία Μαντελή επισήμανε ότι οι δυσκολίες του χρονοδιογράμματος ε, οφείλονται σε μια αλλαγή της στρατηγικής σε ένα δισταγμό που έδειξε αρχικά η Επιτροπή Πολιτισμού προς την ακολουθητέα στρατηγική. Εξού και η σπουδή των τελευταίων ε, ημερών. Και ευχαριστώ θερμά και την εισηγήτρια που εργάστηκε άοκνα και μάλιστα μόνο με μια γλώσσα, τα αγγλικά, αλλά κατέληξε σε αποτελέσματα που πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμα για την ουσιαστική εξέταση αυτού του θέματος και από την Αρμόδια Καθήλια Επιτροπή, που είναι η Επιτροπή Πολιτισμού. Εμείς θα ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση αύριο, τι τροπολογίες δηλαδή τη κυρία Χάρκιν και, της, και η Επιτροπή Πολιτισμού που είναι κατ' ουσίαν αρμόδια, όπως είπαμε, θα ψηφίσει στις 23 Νοεμβρίου μετά από συζήτηση της έκθεσης που θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών στην Επιτροπή Προϋπολογισμών λήγει στις 12 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το σημερινό χρονοδιάγραμμα. Αλλά μερικές φορές τα πράγματα αλλάζουν και δεν είναι αποκρισταλωμένα όπως έχουν αλλάξει τελευταίο καιρό. Αυτά και μια και τελειώσαμε τη μέχρι τώρα ημερή σε διάταξη, είμαι υποχρεωμένη να διακόψω τη συνεδρίασή μας μέχρι τις 5, γιατί τότε θα έρθει ο Επιτρόπος Σαλμούνια. Βέβαια αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, η διακοπή είναι πάντα επικίνδυνη γιατί έχουμε διαρροές σε τέτοιες διακοπές, αλλά σας προσκαλώ να επανέλθετε στην αίθουσα αυτή στι 5 για την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Ευχαριστούμε και τους δήμινες λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Chers collègues, je vous propose de reprendre... Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Σας ζητώ συγγνώμη για την διακοπή που χρειάστηκε να κάνουμε, αλλά υπήρχε έκτακτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το απόγευμα και δεν μπορούσε ο Επίτροπος Αλμούνια να μην παραστεί στη συνεδρίαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το τέλος. Γι' αυτό καθυστέρησε λίγο να έρθει στη δική μας Επιτροπή. Βέβαια είμαστε παλιά γνώριμοι με τον Επίτροπο Αλμούνια και έρχεται εδώ όχι λόγω της προηγούμενης σχέσης που είχαμε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων αλλά για να μας μιλήσει για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την ανάγκη της διάσωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Στις 14 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ε, μετά από πρωτοβουλία και πρόταση του Επιτρόπου Αλμούνια μια ανακοίνωση για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών με μια διάσταση φυσικά και κοινωνική. Οι πρόσφατες τώρα οικονομικές προβλέψεις δημοσιεύτηκαν μόλις σήμερα, οι προβλέψεις για το φθινόπωρο και φυσικά έχουν και μια διάσταση για την απασχόληση που μας ενδιαφέρει άμεσα. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα και θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έρχομαι στην συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχα την ευκαιρία διαλόγου με ορισμένους και ορισμένες από εσά σε μία κοινή συνεδρίαση που είχε γίνει με την Επιτροπή Νομισματικών Θεμάτων υπό την Προεδρία της Περβάνς Μπερές. Και χαίρομαι που δέχτηκα την πρόσκληση της κυρίας Μπερές για να μιλήσουμε για τις ε, οικονομικές προβλέψεις του φθινοπόρου που υπέβαλα χθε και σήμερα το απόγευμα παρουσίασα στο συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ε, θα σας μιλήσω για την ανακοίνωση βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Παρουσίασα στα μέσα Οκτωβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, για τις ε, οικονομικές προβλέψεις του φθινοπόρου. Η χθεσινή μου παρουσίαση είχε τον τίτλο «Η ύφεση τελείωσε». Βγαίνουμε από την ύφεση. Το δεύτερο εξάμεινο του 2009 ήδη δείχνει θετικές ε, τάσεις με βάση όλους τους δείκτες και τους δείκτες δραστηριότητας αλλά και τους δείκτες εμπιστοσύνης και αυτή η βελτίωση άρχισε να γίνεται αισθητή από το δεύτερο τρίμηνο του 2009 και επιβεβαιώθηκε σαφώς στο τρίτο τρίμηνο του 2009. Ευελπιστούμε ότι αυτή η θετική τάση θα διατηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του 2009 αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του 2010. Αυτή βέβαια η θετική πλευρά των προγνωστικών μας συνοδεύεται ή πρέπει να συνοδεύεται από μια εξοενυχιστική ανάλυση κάποιων λιγότερο θετικών πτυχών αλλά και κάποιων ανησυχιών και προβληματισμών για τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης κάποια σχετικά αρνητικά στοιχεία είναι το επίπεδο της ανεργίας. Η ανεργία δυστυχώς αυξάνεται και με βάση τις προβλέψεις μας θα συνεχίσει την ανοδό κατά τη διάρκεια του 2010 και μάλιστα σε συνολικά ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε αύξηση της ανεργίας που θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τη διάρκεια του 2011. και είδαμε ότι και αρχικά αναλύοντας την κρίση αλλά και στην πορεία των οικονομικών μας προβλέψεων διαπιστώσαμε ότι η αρνητική αντίδραση ως προς την ανεργία αλλά και ως προς την απώλεια των θέσεων εργασίας θα γίνονταν αισθητέ με καθυστέρηση δηλαδή μετά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει μία μείωση της απασχόλησης και μάλιστα τα συνολικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ε, κατά 2% αύξηση της απώλειας των θέσεων ε, εργασίας. Και μάλιστα αυτό φαίνεται θα συνεχιστεί και του χρόνου, παρόλο που η ανάπτυξη έχει πια θετικό πρόσημο. Και κατά 2011 για τη ζώνη ευρώ προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί το επίπεδο απασχόλησης, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 προβλέπεται μία μικρή αύξηση της καθαρής απασχόλησης που όμως δεν είναι ακόμη ικανή να απορροφήσει την αύξηση της ανεργίας που προκλήθηκε από την κρίση. Οπότε οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης θα παραταθούν, θα εξακολουθούν να γίνονται και μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με πολιτικές φορολογικών κινήτρων και μακροοικονομικών κινήτρων καθώς και με πολιτικές που θα ενισχύουν την απασχόληση κατά το 2010. Και μόνο το 2011 το γενικό σενάριο ανάπτυξης επιβεβαιωθεί και θα έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε αυτά τα επόμενα τρίμηνα. Μόνο από το 2011 και μετά δικαιολογείται σε συνολικά ποσά μία σταδιακή απόσυρση των κινήτρων. Παρόλο που θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες δραστήριες πολιτικές ενίσχυσης της αγοράς εργασίας, για να γίνουν αισθητέ ε, οι θετικές συνέπειες τη ανάπτυξη και στην απασχόληση. Δεύτερο μειονέκτημα, η αρνητική πτυχή της κρίσης με βάση τη πρόβλεψη, παρά την ανάκτηση τη ανάπτυξης, είναι το επίπεδο του δημόσιου χρέους. Και τα νοικοκυριά και οι οικογένειε, αλλά και οι επιχειρήσει. διανύουν μια περίοδο ισοσκελισμού των ισοζυγίων τους και ένα είδος deleveraging των ισολογισμών τους. Το αντίβαρο όμως είναι μια α, κατακόρυφη αύξηση του δημόσιου χρέους. Και αυτό το δημόσιο χρέος, παρά την ανάκαμψη που θα ξεκινήσει το 2010 και θα ενισχυθεί το 2011, αυτό το δημόσιο χρέος δεν πρόκειται να αποσβεστεί, δεν πρόκειται να μειωθεί ούτε καν το 2011 με βάση τις προβλέψεις μας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης τα επόμενα χρόνια που θα περιορίσει, θα συρρυκνώσει το περιθώριο λιγμών για τη χρηματοδότηση κρατικών πολιτικών που θα ενισχύουν την ανάπτυξη και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Το περιθώριο ελιγμών δηλαδή των δημοσίων οικονομικών μετά την κρίση και για λίγα χρόνια ακόμη θα είναι περιορισμένο. Θα υποστεί πίεση εξαιτία της ε, κατακόρυφης αύξησης ε, του δημόσιου χρέους, εξαιτία της ύφεσης και της χρήσης δημόσιων πόρων για τη χρηματοδότηση των κινήτρων. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις οικονομικές μας αναλύσεις. Έχω και ένα σχόλιο για την κατάσταση των οικοκυριών ή των οικογενειακών οικονομιών. Ούτε το 2009, ούτε το 2010, ούτε το 2011 Ε, εκτιμούσαμε τους ε, κινδύνους πληθωρισμού. Φαίνεται ότι πάντως κίνδυνος από πληθωρισμού έχει εξαφανιστεί. Από άποψη πληθωρισμού λοιπόν, το τοπίο είναι μάλλον καθησυχαστικό. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα ωφεληθεί από αυτή την ουσιαστική και ανυπαρξία του πληθωρισμού ή πολύ χαμηλού πληθωρισμού ή πληθωρισμού που βρίσκεται υπό έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι και ως προς την ανάπτυξη και ως προς την απειλή του πληθωρισμού. Πάντως ε, η ανάλυση μας για τους κινδύνους ε, που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το γενικό σενάριο ε, είναι μάλλον θετική. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σταδιακή ανάκαψη και χωρίς πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Πριν από μία τριετία υποβάλαμε την πρώτη μας έκθεση. Τρία χρόνια μετά, όπως είχε αναγγελθεί το 2006, οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τις 27 χώρες μέλη, εκπώνησαν την έκθεση για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνόδευσε την έκθεση αυτή με μια ανακοίνωση που εγκρίναμε στις 14 Οκτωβρίου. Μία έκθεση βέβαια για μακροπρόθεσμες προβλέψεις γίνεται ε, υπό το σενάριο μιας σταθερής πολιτικής. Και όλες αυτές οι τάσεις και όταν μιλούμε για τάσεις ενό έτου ή δύο ετών είναι προβλέψα. Πολλά δε μάλλον όταν μιλούμε για τάσεις που αφορούν 20-30 χρόνια μετά. Όλες αυτές οι προβλέψεις θα διορθωθούν με αποφάσεις οικονομικής πολιτικής ή με αποφάσεις κοινωνικής πολιτικής ή θα διορθωθούν από κάποιες αλλαγές στον περίγυρο. Πάντως είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για να μας δώσουν μία προοπτική και να δούμε τι θα γίνει αν δεν κάνουμε καμία προσπάθεια για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Γιατί έχουμε και τα δημογραφικά στοιχεία, έχουμε και το σημείο αφετηρίας των δημόσιων οικονομικών, έχουμε τις πληροφορίες για τα επίπεδα απασχόλησης, για την ανάπτυξη. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία καταρτίστηκε η έκθεση που καταλήγει στο συμπέρασμα καταλήγει μάλλον σε ορισμένα συμπεράσματα και σε κάποιες προβλέψεις και προβολές που ελπίζω να τραβήξουν την προσοχή σας. Πιστεύω ότι αξίζουν προσοχής. Αυτές οι προβλέψεις ε, δημιούργησαν κάποιες ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια πίεση για ανάληψη δράσης προκειμένου να μην επιβεβαιωθούν οι αρνητικές τάσεις. Φυσικά το πρώτο που κάναμε είναι να συγκρίνουμε τα συμπεράσματα της έκθεσης του 2009 με τα αντίστοιχα της έκθεσης του 2006 και να δούμε ποιες ήταν οι διαφορές αυτά τα τρία χρόνια. Μέσα σε μία τριετία λοιπόν η μεγάλη αλλαγή ήταν η εμφάνιση της κρίσης που ξεκίνησε το 2008. Οπότε η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και η κατάσταση της απασχόλησης είναι πολύ διαφορετική σήμερα από ό,τι το 2006 και δυστυχώς είναι πολύ χειρότερη από το 2006. Τώρα, αν δούμε τις διαφορές ό,τι αφορά τις δημογραφικές προβλέψεις, σε πολλές χώρες ε, οι δημογραφικές προβλέψεις βελτιώνουν τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Και ένας από τους παράγοντες βελτίωσης σε ορισμένες χώρες ε, ήταν η μετανάστευση. Οι μεταναστευτικές ροές σε ορισμένες χώρες σε αυτή την τριετία που πέρασε από το 2006 μέχρι το 2009 προκάλεσαν αλλαγές στις δημογραφικές προβλέψεις που βελτιώνουν την δημογραφική βιωσιμότητα της ε, πληθυσμιακής εξέλιξης. Σε άλλες χώρες οι μεταναστευτικές ροές δεν είναι τόσο αισθητέ, δεν ήταν αρκετά σημαντικές για να μετατρέψουν αυτές τις δημογραφικές προβλέψεις και έτσι οι προβλέψεις ε, δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2006. Μετά από μία τριετία, οι συνέπειες της γύρας του πληθυσμού για τις δημογραφικές ε, προβολές προσωμιώσεις και για την ανάλυση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών δημιούργησαν κάποιες πιέσεις. Δημιουργήθηκαν πιέσεις στις αναλύσεις αυτές γιατί Σίγουρα όσο γερνάει ο πληθυσμό, οι πιέσει προ τα δημόσια οικονομικά είναι μεγαλύτεροι. Και τρία χρόνια μετά είναι μεγαλύτεροι από ό,τι τρία χρόνια πριν. Σε ορισμένες χώρες ε, με τις μεταρρυθμίσεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη βελτίωση της βιωσιμότητας ε, είχαμε κάποια βελτίωση. Σε ό,τι αφορά την κρίση πάντως και τις επιπτώσεις της, οι νέες δημογραφικές ε, προβλέψεις, τα μέτρα που εθετήθηκαν για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, η μετανάστευση και όλα αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πέντε χώρες, πέντε χώρες μέλη, που με βάση την ανάλυση της έκθεσης παρουσιάζουν μια καλή κατάσταση ως προς τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους. Αυτές οι χώρες αποκαλούμε χώρες χαμηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Και αυτές οι χώρες είναι οι τρεις σκανδιναβικές χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σουηδία, Φιλανδία και Δανία. Και οι δύο είναι νέες χώρες, η Βουλγαρία και η Εστονία. Βέβαια, άλλο να έχει κανείς βιωσιμότητα χαμηλού κινδύνου μακροπρόθεσμη και τα δημόσια οικονομικά σε χώρες που έχουν επίπεδο ευημερία υποδειγματικό και από τα, πιο σημαντικά επίπεδα του κόσμου όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες και να τις συγκρίνουμε με νέες χώρες όπως είναι η Βουλγαρία και η Εστονία που έχουν διαφορετικό επίπεδο ευημερία. Βέβαια, όσο περνά τα χρόνια και στο μέτρο που η ευημερία θα φτάσει ε, και μέχρι τη Βουλγαρία και την Εστονία, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Πάντως η ανάλυση λαμβάνει ως σημείο αφετηρίας τον δημόσιο κλάδο και τα συστήματα κοινωνική προστασία που γνωρίζουμε σήμερα. Έχουμε πέντε χώρε λοιπόν που αποκαλούνται χώρε χαμηλού κινδύνου προ τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Έχουμε εννέα χώρε με μέσο κίνδυνο, η Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Πολωνία και η Πορτογαλία. Αυτέ είναι χώρε μεσαίου κινδύνου ω προ τη βιωσιμότητα. Περίπου οι μισέ δηλαδή χώρε τη ζώνη ευρώ μαζί με δύο νέες χώρες, την Ουγγαρία και την Πολωνία, βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη του μεσαίου κινδύνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ε, τα επίπεδα μεσαίου κινδύνου σχετίζονται με δημοσιονομικά ελλείμματα και το επίπεδο του δημόσιου χρέους. Σε άλλες περιπτώσεις βαρύνει περισσότερο στην ανάλυση η εκτίμηση για τη μακροπρόθεσμη συνέπεια της γύρανσης στα δημόσια οικονομικά των χωρών αυτών. Πάντως, χρησιμοποιώντας τους δείκτες βιωσιμότητας της έκθεση, οι χώρες αυτές βρίσκονται στη ζώνη του μεσαίου κινδύνου, αυτές οι εννέα χώρες. Και 13 άλλες χώρες μέλη αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που τη χαρακτηρίζουμε ως μεγαλύτερο κινδύνο. Είναι οι υπόλοιπε χώρες, δεν χρειάζεται να τις κατονομάσω, γιατί αν αφαιρέσετε από τις 27 αυτές που σας προανέφερα, μα μένουν οι 13 μεγάλου κινδύνου. Και 6 από αυτές τις 13 χώρες έχουν το δίκτυ συναγερμού σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών του. και είναι στη χειρότερη κατάσταση και είναι η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία συγγνώμη, πέντε είναι οι χώρες λέει ο κ. Σαλμούνια Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία και Μεγάλη Βρετανία Αυτέ είναι οι πέντε χώρε που έχουν το δίκτυ στο επίπεδο συναγερμού σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους έχει χτυπήσει κόκκινο για τις χώρες αυτές με βάση τους δείκτες. Τι συνέβη μέσα σε μία τριετία. Πώς ε, εξελίχθηκαν οι χώρες σε αυτή τη σχετική κατανομή σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο βιωσιμότητας. Δέκα χώρες μέλη βρέθηκαν σε χειρότερη θέση από ό,τι πριν από μία τριετία. Και δύο χώρες μέλη, χάρη στις μεταρρυθμίσεις που ε, εφάρμοσαν από το 2006 και μετά, βελτίωσαν τη θέση τους παρά την κρίση και παρά τις συνέπειες της κρίσης. Και οι δύο αυτές χώρες είναι η Ουγγαρία και η Πορτογαλία που παρά την κρίση βελτίωσαν τη θέση τους χάρη στις μεταρρυθμίσεις που θέσπισαν. Και αυτή η ανάλυση αφορά σταθερές πολιτικές δηλαδή αυτό που αναφέρεται ως δείκτης κινδύνου υψηλότερο από το μέσο όρο, δεν σημαίνει ότι ο, κίνδυνος αυτός θα υλοποιηθεί, γιατί με την εφαρμογή των κατάλληλων αποφάσεων είδαμε ότι ακόμη και σε δύσκολες στιγμές όπως είναι η κρίση της τελευταίας, των τελευταίων ετών, ορισμένες χώρες κατάφεραν χάρη στις μεταρρυθμίσεις να βελτιώσουν τους δείκτες βιωσιμότητάς τους. Τις στρατηγικές θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε σε κάθε χώρα. Και οι προτεραιότητες δεν μπορεί να έχουν γενικό χαρακτήρα, ούτε θα πρέπει να έχουμε τέτοιες γενικές προτεραιότητες. Πριν από πολλά χρόνια και πριν τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης το 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χάραξε μια στρατηγική που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη για όλες τις χώρες, όποια και είναι η κατάστασή τους, και αυτή η στρατηγική χωρίζεται σε τρεις ομάδες λύσεων. Η πρώτη λύση είναι να ακολουθηθούν στρατηγικές ε, διόρθωσης των διαρθρωτικών ανισορροπιών των δημόσιων οικονομικών με μεσοπρόθεσμη προοπτική και αυτό βελτιώνει τη βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα στα δημόσια οικονομικά. Δεύτερη προφανής λύση, όσο αυξάνεται η απασχόληση όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τόσο μικρότερη θα είναι ε, και όσο μικρότερη είναι η διαφορά απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών, όσο λιγότερη διάκριση εφαρμόζεται κατά των νέων για την ε, είσοδο και παραμονή της στην αγορά εργασίας, όσο υψηλότερη είναι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας του εργατικού δυναμικού άνω των 50 ετών, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα βελτιώσουν το ποσοστό της απασχόλησης και η βελτίωση του ποσοστού της απασχόλησης βελτιώνει αυτόματα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Και η τρίτη κατηγορία λύσεων είναι κάποιες μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση αυτής της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας με διασταλτική έννοια. Δηλαδή όχι μόνο των συνταξιδοτικών συστημάτων, αλλά και των υπόλοιπων κοινωνικών δαπανών που σχετίζονται με τη γύραση του πληθυσμού ή που κυμαίνονται ανάλογα με την πίεση που επιβάλλει η γύραση του πληθυσμού στα συστήματα κοινωνικής προστασίας ή στα συνταξιδοτικά συστήματα ή στα συστήματα υγειονομικής προστασίας και περίθαλψης. Αυτά, αυτές οι τρεις ομάδες για τη βελτίωση της διάρθρωσης, για την αύξηση της απασχόλησης και για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι κατηγορίες ε, λύσεων που επέτρεψαν σε πολλές χώρες να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις χώρες για να επιτύχουν αυτό το στόχο. Αυτό είναι το συμπέρασμα, το πρωταρχικό συμπέρασμα της έκθεσης. Και αυτή την έκθεση θέλουμε να τη λάβουμε υπόψη για να βελτιώσουμε την ποιότητα των συστάσεων που υποβάλλουμε στα κράτη-μέλη και για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά και για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε στρατηγική της Λισαβόνας και που σύντομα θα αλλάξει όνομα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ήταν σαφέστατα αυτά που μας είπατε. Παρουσιάσατε μια πρόκληση για μας τους πολιτικούς υπεύθυνους που είμαστε. Για την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκουμε, ανεξάρτητα από την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκουμε, έχω μακροσκελή κατάλογο αγορητών που επιμηκύνεται ανάλογα με το που στρέφω το βλέμμα μου, προστίθεται. Λοιπόν, παρακαλώ να είσαστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Παρακαλώ να περιεριστείτε σε τρία λεπτά ο καθένας και έτσι ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους. Θα ακολουθήσω τη σειρά των ε, εγγεγραμμένων, εκείνων δηλαδή που πρώτοι ζήτησαν το λόγο, χωρίς να κάνουμε ιεράρχηση. Κυρία Λίν, ας δώσετε το καλό παράδειγμα παρακαλώ. Και μετά ο κύριος Λέγιαρεκ. Ε, κυρία Λίν, ευχαριστώ, θα κάνω ό,τι μπορώ. Οι δείκτε δείχνουν ότι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε κάποιε χώρε και έχουμε αισθητικά μηνύματα για τον ΑΕΠ. Τι κάνετε όμω σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε να φροντίζετε για δημιουργίε θέσεων απασχόλησης. Ε, διότι είπατε ότι υπάρχει μείωση στην απασχόληση. Και να μην ξεχνούν τα κράτη-μέλη επίση τι ευθύνε του, για να προστατεύσουν του πλέον ευάλωτου από τι συνέπειε της κρίσης. Μπορείτε να αναφερθείτε κάπως στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενθαρρύνει την παροχή πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 37% εκείνων που ρωτήθηκαν σε μια βολιτοσκόπηση που έγινε Γενική Διεύθυνση Αρμόδια για τον ανταγωνισμό είπαν ότι είναι, σε αυτό το ποσοστό είναι πρώτη στην προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Πατρίκ Λεγιαρίκ πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είπατε και σωστά ότι η ανεργία δεν προσθέσατε ότι και η φτώχεια αυξάνεται. Πέραν αυτού, τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξάνονται καθώς και χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Τι μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει άλλη κατανομή του πλούτου όσον αφορά τα δημοσιονομικά. Αυξάνεται το χρέος, τα δημοσιονομικά σε πολλές χώρες είναι στο κόκκινο διότι δώσαν χρήματα στις επιχειρήσεις αλλά μειώνονται κυρίως οι φόροι για τους πιο πλούσιους. Και εσείς μας εξηγήσατε ότι για να ξαναμπεί η οικονομία στο πράσινο πρέπει να μειωθεί το επίπεδο της κοινωνικής προστασίας και το επίπεδο των κοινωνικών δαπανών. Διακόπτει και ο Σαλμούνια, εκεί το είπα εγώ. Είπατε ότι πρέπει να επαναξεταστεί το σύστημα κοινωνικής προστασίας και η διάρκεια ε, θα παραταθεί ο χρόνος ε, συνταξιοδότησης. Δεν αναφερθήκατε στη διαφορά στην ισοτιμία δουλαρίου που είναι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη. Τι θα κάνετε, για να το διορθώσετε. Ξέρω ότι δεν προβλέπετε στο καταστατικό, θα δοθούν όμω προ ανατολισμοί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτω ώστε να ευνοήσει την απασχόληση και όχι την κερδοσκοπία. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση, η κυρία Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, διάβασα προσεκτικά την ανακοίνωσή σας και βρήκα ενδιαφέροντα σημεία. Και στην παρουσίασή σας είπατε ότι η οικονομική εξυγίανση περνά μέσω νέων εσόδων και λέτε ότι η κερδοσκοπία επιβραδύνει την κατάσταση όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και τέλος, υπογραμμίζατε την σημασία να υποστηρίξουμε τα έσοδα των πλέον ασθενών πολιτών μας με διτό στόχο, κοινωνική συνοχή και τόνωση της ζήτησης. Σαν οικολόγος, εγώ συμμερίζομαι τη μεριμνά σας για τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το έλλειμμα σήμερα πληρώνεται από τις μελλοντικέ γενιές, το σημερινό έλλειμμα αλλά να προχωρήσουμε πιο πέρα στην όλη ανάλυση. Το Δεκέμβριο του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε μια σύσταση για να πλησιωθεί ε, το πλαίσιο, να θεθούν όρια στα όρια των υψηλών στελεχών. Τόσα χρόνια μετά δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Η σύσταση εν μέρη εφαρμόστηκε και κάθε ειδών καταχρήσει αυξήθηκαν. Το bonus, το stock auction, η πρόορη συνταξιοδότηση. Κάθε χρόνο, κύριε Επίτροπε, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα μοιράζονται πιο πλούσιοι. Ενώ οι φτωχότεροι, που είναι οι εργάτε, οι εργαζόμενοι κλπ., βλέπουν απειλείται η δουλειά του από τι μετεγκαταστάσει των επιχειρήσεων και από την κερδοσκοπία όσον αφορά τι χρηματοδοτικέ αγορέ και ότι μένουν σταθεροί και μειώνονται οι μισθοί του λόγω του πληθωρισμού. Θα έλεγα ότι οι διαφορέ των εισοδημάτων πήγαν από 1 στο 10 στη δεκαετία 70 είναι 1 προς 60 τώρα, ενώ ήταν 1 προς 10 τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έκανε μια πρόταση οδηγία που έχει σαν στόχο μεταξύ άλλων μια εποπτεία συνετής διαχείρισης όσον αφορά την πολιτική των αμοιβών, κυρίως στον τομέα των χρηματοστοτικών υπηρεσιών. Είναι κάτι αναγκαίο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά, διότι σήμερα αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει σήμερα να προχωρήσουμε πιο πέρα όσον αφορά τα πλαίσια των υψηλών αμοιβών και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μια φορολογία που θα περιορίζει τα πολύ ψηλά εισοδήματα, περιορίζοντας το 90% όλα τα εισοδήματα που είναι πάνω από, τα, από 30 φορές το μέσο μισθό. Και έτσι θα ρυθμιστεί το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων. Το 1942 το έκανε ο Ρούσβελτ και αυτό κάνει σήμερα και ο πρόεδρος Ομπάμα. Έτσι θα είχαμε μια νέα πηγή φορολογικών εσόδων που θα επέτρεπε να συμμετάσχουμε έτσι στην εξυγίανση των δημοσιονομικών και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της κερδοσκοπίας στην πραγματική οικονομία. Και τα νέα έσοδα θα επιτρέψουν την ενίσχυση του συστήματος προστασίας και θα εγγυηθούμε ένα ελάχιστο εισόδημα για όλου. Και του συνταξιούχου, για του σπουδαστέ, για του ανέργου, του φτωχού εργαζομένου. Θα ήθελα να ξέρω συγκεκριμένα τι θα προτείνετε λοιπόν για να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με ακρίβεια αλλά και λακωνικότητα. Καταρχήν, ως προς την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Φυσικά, πολλά θα πρέπει να γίνουν για τους λόγους που σας εξήγησα και προηγουμένως. Γιατί αν δεν δράσουμε, αν δεν αναλάβουμε δράση για να βελτιώσουμε την ικανότητα των οικονομιών μας, για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, εφόσον ήδη υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης, θα αντιμετωπίσουμε όχι μόνο υψηλή ανεργία βραχυπρόθεσμα, αλλά και διαρθρωτική μακροπρόθεσμη ανεργία. Κάτι που θα κρατήσει εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία, ακόμη και με οικονομική ανάκαμψη ή ανάπτυξη, κάτι που θα πρέπει να αποφευθεί οπωσδήποτε. Και επίσης θα έχουμε διασπάθηση ανθρωπίνων πόρων, γιατί το τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό μένει αναξιοποίητο. Κάτι που συρρυκνώνει τη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν οι εθνικές αρχές, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί φορείς ε, σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προβούν σε μια κατεπίγουσα και πολύ εμβριθή ανάλυση πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, ή τι μέτρα θα πρέπει να λάβουν για να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να ενισχύσουν την απασχόληση. Μάλιστα θα αρχίσει τους επόμενους μήνες μία συζήτηση για τις ε, μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Κάτι που θα ενισχύσει αυτή την ευρυθή συζήτηση. Βέβαια, η εύκολη απάντηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα σχήρας της δεν έχει σχετικές αρμοδιότητες, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει ε, προϋποθέσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης. Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις, δεν το ανέφερα, αλλά η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές λειτουργούν πια πιο ομαλά από τη στιγμή της κρίσης, γιατί τότε διατρέχαμε τον κίνδυνο μιας ε, πλήρους κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή όμως η εξομάλυνση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών δεν οδήγησε αυτόματα σε ανάκαμψη της πίστοσης. Οι ροές της πίστοσης ε, προς οικογένειες κυρίως και προς μη κερδοφόρες επιχειρήσεις ε, βρίσκονται σε μηδενικό επίπεδο και χωρίς τέτοια ροή δανείων δεν θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν οι οικογένειες και οι ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό από την αρχή της κρίσης ενισχύσαμε τα προγράμματα στήριξης με τους διαθέσιμους πόρους που είχαμε σε κοινοτικό επίπεδο προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρησιμοποιώντας πόρους από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και μέσω του προγράμματος SIP και με δράσεις της Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, αλλά και με, σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικές χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των, Ευρωπαϊ... χωρών μελών προσπάθησαν να βελτιώσουν τις χρηματοληπτικές πιστοληπτικές ικανότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βέβαια όλα αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια δανεισμού από τις χρηματοπιστωτικές μονάδες. Κάτι που είναι απαραίτητο να διορθωθεί. Θα πρέπει να γίνει μια ανάκαμψη των πιστώσεων που θα παρέχονται και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και σίγουρα η ανάκαμψη σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διονύσει τις ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν από το προηγούμενο σύστημα που μας οδήγησε στην κρίση. Γιατί λόγω της αδικίας που επικράτησε αυξήθηκαν οι ανισορροπίες. Και η κρίση προκάλεσε όχι μόνο ένα προβληματισμό για τα θέματα αυτά, αλλά και ένα είδος δυσανεξίας της κοινή γνώμης σε ό,τι αφορά την διαιώνιση τέτοιων ανισορροπιών και ανισοτήτων σαν αυτές που είχαμε πριν από την κρίση. Ο κόσμος πια δεν ανέχεται μια παράταση αυτής της κατάστασης ανισορροπίας. Και σίγουρα τα φορολογικά συστήματα θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν μπορούν ε, τα φορολογικά συστήματα να προβούν σε ανακατανομή του πλούτου και σε διόρθωση των ε, ανισοτήτων. Θα πρέπει πέραν των φορολογικών ε, κινήτρων να χρησιμοποιηθούν και άλλοι μηχανισμοί από την πλευρά των δαπανών του προπολογισμού. Επίσης, να χρησιμοποιηθούν κάποιοι μηχανισμοί για την ενίσχυση κάποιων δραστηριοτήτων και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης ε, για κλάδους που είχαν διαφύγει του ελέγχου και της ρύθμισης τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε από αυτή την άποψη την κρίση, να μην πάει χαμένη ως προς τη βελτίωση της ρύθμισης. Και θα πρέπει σε συνεργασία, με συνεργασία όλων των αρχών και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων να διδαχθούμε από αυτή την κρίση και να την αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε. Γίνεται μια προσπάθεια, αλλά φυσικά δεν έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες, θα πρέπει να συνεχιστούν. Το σχόλιο σας ε, για την περικοπή συρρήκνωση των κοινωνικών δαπανών είναι τελείως άσχετο με αυτά που είπα. Εγώ μίλησα για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και η βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας δεν έχει καμία σχέση με τη συρρήκνωση των κοινωνικών δαπανών. Θα πρέπει όμως να εγγυηθούμε στις επερχόμενες γενιές τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο κοινωνικών δαπανών που απολαμβάνουμε εμείς. Δεν ξέρω τι μου δείχνετε γιατί δεν μπορώ να διαβάσω από τέτοια απόσταση. Φέρτε το μου διαβάστε το μου αν θέλετε να το καταλάβω. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη περικοπής των κοινωνικών δαπανών για να βελτιώσουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Το αντίθετο, αν δεν βελτιωθεί η βιωσιμότητα, αποκλείεται να διατηρηθούν να παραμείνουν βιώσιμα αυτά τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Και αυτός είναι ένας πραγματικός κίνδυνος που θα πρέπει να τον λάβουμε υπόψη. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα νέων εσόδων ή νέων φόρων, σίγουρα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση και ένα τμήμα των εσόδων χρηματοδότησε την κρατική δραστηριότητα πριν από την κρίση και δεν θα χρησιμοποιηθούν μετά την κρίση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέες φορολογικές βάσεις που θα αντικαταστήσουν τις προηγούμενες και φυσικά έχουμε κάποιους φόρους που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα το περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτή είναι μία ίσως από τις πηγές ε, φορολογικών εσόδων που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αναδιανεμητικά συστήματα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και τον ιδιωτικό κλάδο. Η ανάλυση της κρίσης μας επέτρεψε όχι μόνο να κάνουμε κάποιες ε, σκέψεις ιδεοντολογικές και ηθικές ό,τι αφορά την αναδημητική δικαιοσύνη με βάση ένα σύστημα αντιστάθμισης αλλά υπάρχει συνένεση σε επίπεδο G20 τουλάχιστον ότι αυτά τα συστήματα τα διανεμητικά δημιούργησαν ακριβώς τα κίνητρα που οδήγησαν την γέννηση της κρίσης. Γιατί δημιούργησαν κίνητρα προκυκλικά, προσυγκυριακά, οδηγήσαν στην ανάληψη παράλογων κινδύνων. Τώρα καλός ή κακός δεν μπορούμε να θεσπίσουμε κάποιες, κάποιους κανόνες μέσω οδηγιών. Ούτε εσείς ούτε εμείς έχουμε αρμοδιότητες για την επιβολή μέτρων, αλλά στο μέτρο που μπορούμε να έχουμε συζήτηση και να εξηγήσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτών των διανεμητικών συστημάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πυθό για να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας απομένει κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Έχω 16 εγγεγραμμένους και κλείνω τον κατάλογο. Και ζητώ από καθένα από εσά να μιλήσετε για ένα λεπτό. Η κυρία Ράπτη και ο κ. Μπούλμα μετά. Η κυρία Ράπτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον κύριο Αλμούνια και θα χρειαστώ λιγότερο από ένα λεπτό. Προέρχομαι από μία από τις πέντε χώρες που είναι στο κόκκινο. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι στο νότο, έχουν απόκληση από το κοινωνικό και εκτιμένο σε σχέση με τα κοινωνικά συστήματα υγείας και με αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, γιατί, ζητούν, γιατί ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπουν οι ίδιοι φόροι και σε αυτά τα κράτη, μερικά από τα οποία κάνουν προσπάθεια να κερδίσουν το χαμένα έδαφος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ότε Ο κύριος Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν να αντιδράσουν στην αυξανόμενη ενεργεία μειώνοντας, ε, κρατώντας μάλλον τους υπαλλήλους τους με χαμηλότερο, μικρότερο ωράριο ή συνοδεύοντας τους ανέργους προκειμένου να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας και πληρώνουν ε, υψηλούς ε, μισθούς υποκατάσταση. Δηλαδή θέλουν να αναπτύξουν γρήγορα το απόθεμα αυτών των εργαζομένων. Από τη δική σας ε, πλευράς δεν θεωρείτε ότι αυτή τη στρατηγική θα έπρεπε να την υποστηρίξουμε, δεν θα, υπάρξει, δεν θα έπρεπε να υπάρξει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να το ακολουθήσουν όλοι αυτό το πρόγραμμα. Δεν θα πρέπει να τεθούν benchmarks για τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα, προσπαθούσαμε, δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τα προγράμματα αυτά από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. ευχαριστώ πολύ. Και μετά ο κ. Πουπάκης. Euh, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της λέει ότι μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους δεν μπορεί να υπονομεύει τα δημοσιονομικά, τη βασιμότητα δημοσιονομικά. Δεν μπορεί να τα θέσει κίνδυνο θα έλεγα. Γιατί είναι γενικόλογη διατύπωση, θα μπορούσε να πει συγκεκριμένη και λέτε υπερβολική συσσόρευση δημόσιου χρέους με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο και υπονόμευση των δημοσιονομικών και στις πρόσφατες εξελίξεις υποτίθεται ότι στην Ευρωζώνη θα πλησιάσουμε το 2011 οικονομικό χρέος περίπου 100% του ΑΕΠ είναι κάτι που μπορούμε να το χειριστούμε είναι υπερβολικό έχοντας υπόψη ότι στις χώρες όπου τέτοια χρέη υπήρχαν κατά το παρελθόν και ότι αυτό επιφέρει επιβάρυνση ενός τετάρτου ε, ε, του, του δημοσίου χρέους για την επόμενη γενιά. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και συμπληρωματικές δαπάνες που που σχετίζονται με την αυξανόμενη ανεργία στο Λουξεμβούργο, στη χώρα μου και μόνο. Το Ταμείο για την Απασχόληση που πληρώνει το επίδομα ανεργίας αύξησε τις δαπάνες κατά 100%. Διπλασιαστήκαν οι δαπάνες. Από μισό εκατομμύριο, δισεκατομμύριο ευρώ φτάσαμε στο ένα δις ευρώ τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ, διακόπτη η Πρόεδρο. Μιλήσατε σχεδόν διπλάσιο από το χρόνο σα. Ο κ. Πουπάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την παρουσία σα, κύριε Επίτροπε. Θέλω να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντική την επισήμανση τη Επιτροπή για την αναγκαία διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών για να μειωθεί το χάσμα βιωσιμότητα, όπου η όποια μεταρρύθμιση να μην διευρύνει ή να πολλαπλασιάζει τι επιπτώσει οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Όπω για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί να μειώνονται οι συντάξει όταν επιβάλλεται αυξημένη αγοραστική δύναμη των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων για την αντιμετώπιση τη ύφεση. Παρά λοιπόν αυτό το επιβεβλημένο, όπου τα δημόσια οικονομικά σαν σύνθετο μέγεθο θα συνεξετάζονται στο πλαίσιο τη συνολική οικονομική και κοινωνική πολιτική, έχω την αίσθηση ότι παραλείπονται συχνά, ίσω και συστηματικά. Θα ήθελα λοιπόν καταλήγοντα να ρωτήσω σε αυτή τη δύσκολη ακόμα περίοδο τη κρίση για τι ανισότητε που κι εσεί αναφέρατε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στην πρόθεση της να προτείνει κάποια πιο συγκεκριμένα μέτρα μέσα από μια πολιτική διαχείρισης δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο μιας γενικευμένης αναδιανομής του εισοδήματος προς όφελος των οικονομικά στενέστερων κοινοτάξεων, χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων, δηλαδή φτωχών εργαζομένων και ανέργων. Και αν μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και μέτρα για την ένταξη των οικονομικών μεταναστών. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με την ίδια ταχύτητα. Ως προς την πρώτη παρατήρηση, όταν οι εθνικές οικονομίες ή οι περιφερειακές οικονομίες στην παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζουν κάποιες ανισορροπίες, θα πρέπει αυτές οι ανισορροπίες να διορθωθούν για να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό απαιτεί κάποιες ε, ρυθμίσεις και προσαρμογές. Και όταν γίνονται τέτοιες ρυθμίσεις κάποιος θα χάσει αυτά που είχε. Γιατί δεν μπορεί να γίνει προσαρμογή με τελείως ανώδυνο τρόπο. Και τώρα στους χαλεπούς καιρούς πώς θα γίνει η κατανομή των θυσιών αυτής της προσαρμογής και σε, στην περίπτωση ανάπτυξη, στην περίοδο της ανάπτυξης των παχιών αγελάδων πώς θα διανέμονται τα κέρδη και τα ωφέλη σε μια εύρωστη οικονομία. Μια οικονομία που δεν είναι ανταγωνιστική μια οικονομία που δεν έχει την ικανότητα ανταγωνισμού σε μια ανοιχτή αγορά, γιατί δεν διαθέτει αρκετή σώρευση κεφαλαίου, δεν διαθέτει αρκετή δίκευση ανθρώπινου δυναμικού, δεν διαθέτει αρκετή τεχνολογία, μια τέτοια οικονομία δεν μπορεί να δημιουργήσει να παράγει το ίδιο πλεόνασμα για να το διανύμει μεταξύ των πολιτών της, όπως μια εύρωστη οικονομία, μια ισχυρή οικονομία και ακμαία που έχει σωρεύσει πλούτο, έχει σωρεύσει κεφάλαιο και έχει ένα πλεόνασμα η απόθεμα και ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου και διαρθρώσεων για χρόνια ολόκληρα. Από άποψη οικονομικού ορθολογισμού αλλά και πολιτικού ορθολογισμού δεν μπορούμε να περιμένουμε μια χώρα με 10.000 ευρώ να εξασφαλίσει το ίδιο ποσοστό ευημερία αντίστοιχη με μια χώρα που έχει κατακεφαλήν εισόδημα 30.000 ευρώ. Οι οικονομίες πάντως που έχουν ένα επίπεδο ευημερία πολύ σημαντικό και πολύ αποτελεσματικό και πολύ πιο δίκαιο στην Ευρώπη είναι οι οικονομίες που δεν καταβάλουν οικονομικό τίμημα για την ευημερία τους αυτή αλλά κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια σωστή συνεργασία μεταξύ πλούτου και ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής προστασίας και μείωσης των ανισορροπιών και των ανισοτήτων. Αυτό είναι το κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο. Βέβαια δεν βρίσκονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στο ίδιο επίπεδο, αλλά όλοι συμφωνούμε ως προς το ιδεατό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Ούντο Μπούλμαν. Στο τελευταίο άτυπο εκοφήν, και στο επόμενο εκοφή που θα γίνει την Τρίτη θα συζητήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ό,τι αφορά τις αγορές εργασίας. Γιατί αυτό το θέμα προβληματίζει όχι μόνο τους Υπουργούς Απασχόλησης και ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και αυτό το ξέρετε γιατί είστε μέλη αυτής της Επιτροπής και έχετε συνομιλίες με τους αρμόδιους Επιτροπής και του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά αλλά και στο ΕΚΟΦΗΝ και εγώ ως Επίτροπος Οικονομίας ανησυχούμε για τα θέματα της απασχόλησης. Και μάλιστα στο Γκέτεμπορκ, στο άτυπο συμβούλιο του προηγούμενου μήνα, αλλά και την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, θα εξετάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές των πολιτικών ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ε, θέματα κινητικότητας εσωτερικής, ε, ελαστικότητας, flexicurity, χρήση των πόρων για τις πολιτικές απασχόλησης και πολιτικές καταπολέμησης ανεργίας. Θα δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές ώστε να έχουμε στην απασχόληση τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο συντομότερο δυνατό διάστημα. Γιατί αυτά τα θέματα απασχολούν όχι μόνο του υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και απασχόληση, αλλά και του ε, ηθήνοντε για οικονομικά θέματα. Θέλουμε μια άμεση ανάκαμψη και των επιπέδων απασχόληση, σε επίπεδα που είχαμε πριν την κρίση. Αλλιώ δεν μπορούμε να μιλούμε για έξοδο, βιώσιμη έξοδο από την κρίση αν δεν αποκαταστήσουμε τα παλιά επίπεδα απασχόληση. Αυτή η συζήτηση είναι απαραίτητη. Και εκεί το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει από κοινού να σκεφτούν πώ θα αξιοποιήσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα κονδύλια του κοινοτικού προπολογισμού και κυρίω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά υπάρχει ένα σαφέ περιθώριο και ευρύ περιθώριο για να βελτιωθεί, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των πόρων. Κύριε Έγκερ, συμφωνώ ότι το υπερβολικό δημόσιο χρέος συνεπιφέρει πολλά προβλήματα. Βραχυπρόθεσμα είναι αναπόφευκτη αύξηση του δημόσιου χρέους και είναι αναπόφευκτη η αύξηση με το ρυθμό, το ραγδαίο ρυθμό που επιτελείται, αλλά Ξέρουμε ότι θα πρέπει ήδη να χαράξουμε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση και να αποσβέσουμε ή να μειώσουμε το δημόσιο χρέος ή το πλεόνασμα δημόσιου χρέους που δημιουργήθηκε από την κρίση. Γιατί σε ορισμένες χώρες αυξήθηκε κατακόρυφα ε, η να μειωσουμε το δημοσιο χρεος το χρέωση, αλλά προσπάθησε να, οι χώρες αυτές να προβούν σε μια εξυγίαση των οικονομικών τους και άλλες χώρες, χωρίς να έχουν εξηγιάνει την προηγούμενη τους οικονομική κατάσταση, συνέχισαν να αυξάνουν το δημόσιο τους χρέος. Αυτές οι χώρες θα χρειαστεί να κάνουν πολύ περισσότερες προσπάθειες. Αλλά προσπάθειες θα χρειαστούν όχι μόνο επειδή έχουμε υψηλό δημόσιο χρέος, αλλά επειδή η ανάπτυξη των επόμενων χρόνων θα είναι μικρότερη από την ανάπτυξη πριν την κρίση. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τα θεμέλια μιας μεγαλύτερης ανάπτυξης γιατί και η ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι πολύ μικρότερη από ό,τι αυτή που είχαμε πριν την κρίση. Γιατί αρχικά είχαμε και προϋπολογισμό 2, 2,5, 3%, ενώ σήμερα ο πληθωρισμός είναι μεταξύ 0 και 1 στις περισσότερες χώρες τα 100. Οπότε και εκεί η αναλογία δημόσιου χρέους ΑΕΠ μειώνεται ενώ η αναλογία δημόσιου χρέου, ΑΕΠ αυξάνεται. Όχι επειδή αυξάνεται, αλλάζει ο δείκτης, το δημόσιο χρέο, αλλά και ε, το μέγεθος που χρησιμοποιείται για να ληφθεί υπόψη η εκτίμηση αυτού του δημόσιου χρέου. Τώρα, αν κατάλαβα καλά αυτά που είπε ο κύριος Πουπάκης, θα πρέπει να δούμε ποια, ποιες είναι οι μελλοντικές μας δεσμεύσεις για τα κοινωνικά θέματα, για τα θέματα υγείας και ούτω καθεξής. Ο διευθυντής ε, του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου υπέβαλε ε, το προηγούμενο μήνα στην Κωνσταντινούπολη μια γραφική παράσταση που είναι πολύ χαρακτηριστική. Είχε σε μια στήλη τις μελλοντικές δεσμεύσεις που ήδη αναλάβαμε στη διάρκεια της κρίσης για να υποστηρίξουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα με σημαντικές ε, προτάσει σε απόλυτου όρου και δίπλα είχε τι μελλοντικέ δεσμεύσει που ανέλαβαν οι χώρε μα για να ικανοποιήσουν τι ανάγκε σύνταξη αυτή τη γενιά, αλλά και των μελλοντικών γενιών δεσμεύσει που ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούνται οι ανάγκε νέων εργαζομένων που αρχίζουν και δημιουργούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα για το μέλλον. Και οι παράγωγε δεσμεύσει από τι συνέπειε τη γύρα του πληθυσμού είναι πολύ μεγαλύτερε από τι δεσμεύσει που δημιουργήθηκαν για την υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και μάλιστα οι δεσμεύσει ε, που αναλύθηκαν για, το, για τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν πολύ μεγάλες. Αλλά για, τις, ε, για την εξασφάλιση των συντάξεων ήταν ακόμη μεγαλύτερες αυτές οι δεσμεύσεις. Και ήδη από τώρα θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη βιωσιμότητα αυτής της προστασίας αν θέλουμε πραγματικά να εγγυηθούμε αυτή την προστασία και στις επερχόμενες γενιές. Ευχαριστώ κύριο Σανταμ Κώσα έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το ερώτημά μου αφορά τα άτομα με αναπηρίες. Πριν από δύο εβδομάδες έθεσα ερώτημα στον Πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα και θέλω να θέσω πιο συγκεκριμένο ερώτημα επ' αυτή τη ευκαιρία. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οι εργαζόμενοι με αναπηρία στηρίζονται από την κυβέρνηση. Οπότε στον τόπο εργασίας υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Υπάρχει νόμος που το εγγυάται αυτό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικός στόχος. Δυστυχώς λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσεως όμως έγιναν περικοπές στην στήριξη προς αυτά τα άτομα στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και πολλοί άνθρωποι με αναπηρία έχασαν τη θέση τους την εργασία τους εξαιτία αυτού. Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηριχθούν αυτοί οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, αυτοί που δεν φταίνε για την κρίση και αυτοί δέχονται τις συνέπειες της κρίσης περισσότερο κατά το παρελθόν. Μάλλον δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε περικοπές σε αυτό το τομέα. Λίμπια Κοτσάρη, και μετά η κυρία Λίζα Μόραν. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω το εξή ήθελα. Έχετε εμπιστοσύνη στα μοντέλα με τα οποία ε, γίνεται μέτρηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της ε, ικανότητάς τους έχω τις αμφιβολίες μου. Λαμβάνεται για παράδειγμα υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει χρέωση παράλληλα με την αύξηση της ε, ανεργίας ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, αλλαγές στην οικονομία, στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε πολλές ε, βιομηχανίες, γύρανση του πληθυσμού, όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση. Είπατε ότι για παράδειγμα στη χώρα μου τα πράγματα βρίσκονται υπό έλεγχο. Αλλά και σε μας υπάρχει τάση επιδείνωσης. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ο κόσμος βγαίνει πιο νωρίς ε, στη σύνταξη. Μειώνεται δηλαδή ο χρόνος, ε, υπηρέτητας εργασίας. Τα έχετε λάβει όλα αυτά υπόψη. Σε ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ελίζαμπεθ Μόργαν και μετά η κυρία Ήλτα Φιγκερείδο. Κύριε Επίτροπε, διάβασα με μεγάλη προσοχή την ανακοίνωσή σας και σας άκουσα και έχω τρεις παρατηρήσεις και ερωτήσεις να σας θέσω. Και εγώ διαιρωτώ με όσον αφορά αυτό το μοντέλο. Και το πρώτο ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου. Διερωτώ με σήμερα με το σύστημα υγείας ανεξάρτητα από το πρόβλημα της γύρανσης που θίξατε. Σκέφτομαι και ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος. Οι, δημόσια, οι δημόσιες πολιτικές ανέπτυξαν πολιτικές εντοπισμού του καρκίνου και πρέπει να ληφθούν υπόψη οικονομικές συνέπειες αυτών των πολιτικών. Καμία χώρα όμως, κανένας δεν θα ήθελε να επαναχωρήσει όσον αφορά την οικονομική πολιτική που ακολουθείται εκεί. Δεύτερον, υπογραμμίσατε ότι η παιδεία, η έρευνα και η ανάπτυξη και η καινοτομία είναι μοχλή για το μέλλον, για να βγούμε από τον φαύλο κύκλο αυτό στον οποίο έχουμε κλειστεί. Πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά αυτές τις πολιτικές με περιθώρια οικονομικών ελιγμών πάρα πολύ μικρά. Τρίτον, παρουσιάσατε μια κατάσταση ευρωπαϊκή αλλά τι γίνεται ε, με συσχετισμό της οικονομικής κατάστασης Ευρώπης σε σχέση με την ε, κατάσταση που στην Ινδία, τη Βραζιλία, την Κίνα, την, ε, την, τους αναδιόμενες χώρες. Σήμερα αυτό θα μας δυσχεράνει οικονομικά. Στο μοντέλο σας πώς εισάγεται τις αναδιόμενες οικονομίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ήλντα Φιγερέιδο, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω και εγώ στο θέμα της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Ο Επίτροπος μας είπε ότι παρά την κρίση, πολλές, μερικές χώρες όπως η Πορτογαλία βελτίωσαν την κατάστασή τους. Αν το λέγατε όμως αυτό στην Πορτογαλία, κύριε Επίτροπε, ο κόσμος θα σας πει ότι κάπου λάθος έχει αξιολόγησή σας. Γιατί η ανεργία καλπάζει. Κάθε μέρα κλείνει μία επιχείρηση. Υπάρχει την κατάσταση πολυεθνικών. Η φτώχεια είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που αυξάνεται καθημερινά. Ο πληθυσμός της Πορτογαλίας ζει όλο και χειρότερα. Το βιωτικό επίπεδο μειώνεται. Και μάλιστα θα έχουμε και την πιθανότητα ανακοίνωση για τη μη τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητα. Ενώ ο πληθυσμό, ο κόσμο, οι εργαζόμενοι οι φτωχοί που είναι πάνω από τα 20% του πορτογαλικού πληθυσμού αντιμετωπίζουν συνθήκε πραγματική φτώχεια. Διαρωτάτε λοιπόν ο απλό πολίτη θα, θα επιταθούν τα μέτρα και αντί για 20% φτωχών να φτάσουμε σε 30-40% των φτωχών γιατί θα περιοριστούν τα κέρδη, γιατί οι εργαζόμενοι που σήμερα είναι άνεργοι πολλοί από αυτούς δεν λαμβάνουν καν ε, επίδομα ανεργίας, πάνω από τους μισούς ανέργους δεν έχουν καν ε, επίδομα ανεργίας. Εδώ βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας κοινωνικής τραγωδίας και εσείς μας υπόσχεστε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρέπει να είστε ακόμη πιο επιγραμματικός. Ναι, γρήγορα λέει ο Επίτροπος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ στις Βρυξέλλες ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να, να δείξουμε σε κάθε κάτω μέρο πώ να κάνουν την προσαρμογή των δημοσίων οικονομικών του. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Λέμε ότι αυτό ο προπολογισμό χρειάζεται προσαρμογή λόγω των χρεών που αναφέραμε, βιωσιμότητα, τη δυνατότητα να πληρωθεί, να καλυφθεί το χρέο για κάθε χώρα. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε εν ονόματι των κυβερνήσεων και των εθνικών κοινοβουλίων με ποιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα έσοδα και τις δαπάνες του προϋπολογισμού, θα κινηθούν. Και κάποια κεφάλαια των δαπανών έναντι άλλων, πώς θα κάνουν τη σωστή κατανομή των πόρων και πώς θα κάνουν θυσίες και πώς θα αποκομίσουν ωφέλη από τις προσαρμογές. Όταν υπάρχει δυνατότητα να, να γίνουν οι προσαρμογές αυτές χωρίς με κάποιους όρους ε, προσέχουμε να γίνεται ισότιμα η κατανομή των πόρων. Αλλά όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοχλό όσον αφορά τις πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις που αφορούν το εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε εμείς τις ευθύνες των εθνικών αρχών και την αντιμετώπιση των πληθυσμών, των ατόμων με αναπηρία στις διάφορες χώρες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να αντικαταστήσουμε τις εθνικούς φορείς, τις εθνικές ευθύνες, εκτός από τα επίπεδα εκείνα που επιτρέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που κινηθούμε. Είναι αλήθεια ότι οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ένα επίπεδο υψηλό κοινωνικής προστασίας, έχουν εύρωστα οικονομικά, έχουν εξασφαλίσει ένα επίπεδο ευημερία και έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τους πόρους από τις, εται, από τις εταιρείες τους, τους πολίτες για να χρηματοδοτούν τις προσπάθειές τους. Και είναι αξιοζήλευτες αυτές οι σκανδιναβικές χώρες για τον τρόπο που τα έχουν καταφέρει. Βέβαια και αυτές οι χώρες ε, αντιμετωπίζουν κάποιες αδυναμίες και κινδύνους. Και η κυρία Γιακοσάρη επισήμανε ένα τέτοιο κίνδυνο. Αναφερθήκατε στην πρόοριση δεξιοδότηση. Με την κρίση αυτή σχεδόν όλες οι χώρες διδάχθηκαν από τα παθήματά τους και από τα λάθη τους προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν προηγούμενες κρίσεις. και δεν έχουμε κύμα πρόωρων συνταξιδοτήσεων. Κάτι που στις προηγούμενες κρίσεις οδήγησε ε, στην απόλυση από την αγορά εργασίας, ε, στην αποπομπή από την αγορά εργασίας εργατικού δυναμικού που ήταν 50 ετών ή 55 ετών. Νομίζω ότι αυτό το, το πάθημα μας δίδαξε κάτι. Βέβαια μπορεί να υπάρξουν νέες εκπλήξεις, γιατί μία μελέτη συντάσσεται από εμπειρογνώμονες, όχι από προφήτες. Οι εμπειρογνώμονες δεν είναι προφήτες και δεν είναι προφήτες αυτοί που συντάσσουν εκθέσεις. Απλώς προσπαθούν με τις μελέτες τους να προβάλλουν στο μέλλον την εμπειρία που διαπιστώνουν από το παρόν. Αλλά δεν είναι ε, και προφήτες για να προβλέψουν ε, με ακρίβεια τι θα συμβεί μετά από μία δεκαετία, τι λάθη θα πρέπει να αποφευχθούν από τις ε, κυβερνήσεις ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές οι προσωμιώσεις ή προβλέψεις γίνονται με σταθερή πολιτική. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε λάθη για να τα αποφύγουμε, για να απαλλάξουμε τους ηθήνοντες από την ε, διάπραξη τέτοιων λαθών. Μία τέτοια μελέτη έχει και περιορισμούς, έχει και τα όρια της. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, ε, περιλαμβάνεται και αυτό στην έκθεση. Τώρα, αν υπάρχει περιθώριο για πολιτικές παιδείας, ε, καινοτομίας, τεχνολογικής ανάπτυξης, έρευνας, φυσικά και υπάρχει περιθώριο για τέτοιες πολιτικές και κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία το διατρανώνουμε. Δεν είναι αυτές οι δαπάνες που θα πρέπει να θυσιαστούν για τις δημοσιονομικές προσαρμογές και περικοπές. Γιατί αυτές είναι επενδύσεις και οι χώρες με λιγότερο α, ανισόρροπους προϋπολογισμούς έχουν και μεγαλύτερο περιθώριο. Γι' αυτό και θα πρέπει οι χώρες να ισοσκελίσουν το συντομότερο δυνατό τα δημόσια οικονομικά τους. Σε ό,τι αφορά τώρα την καταπολέμηση της φτώχειας. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε κρατικές πολιτικές, παιδείας, έρευνας, τεχνολογικής και καινοτομίας. Χρειαζόμαστε δημόσιους πόρους για κάτι τέτοιο. Και αν οι προπολογισμοί είναι ανισόρροπη, δεν είναι ισοσκελισμένη, οι πόροι του το προϋπολογισμού θα, θα εξυπηρετήσουν κυρίως την αποπληρωμή του χρέους και δεν θα χρηματοδοτήσουν τέτοιες, τέτοιους σημαντικούς τομείς. Τώρα για τις αναφιόμενες, οικονομίε, οικονομίες, Κίνα, Βραζιλία κτλ. Είναι μια ευκαιρία. Α μην φοβόμαστε αυτέ τι χώρε. Α μην φοβόμαστε αυτέ τι αναδυόμενε οικονομίε. Να χαρούμε για, την θετική τους πορεία και να αξιοποιήσουμε αυτή την θετική εμπειρία που έχουν αυτές οι χώρες που είναι και πολυπληθείς. Γιατί όλοι στον ίδιο κόσμο ζούμε και αν αλληλοϊποστηριχθούμε η βελτίωση θα μας ωφελήσει όλους. Δεν θα πρέπει να ενδώσουμε στο φόβο, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες τις ευκαιρίες που μας δίνει το γεγονό ότι η Κίνα αναπτύσσεται με ρυθμού 8%. Ε, η Ινδία έχει επίσης πολύ σημαντική ανάπτυξη. Η Βραζιλία πάει πολύ καλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αυτά δίνουν ευκαιρίες και σε εμά, γιατί εμείς ε, οι Ευρωπαίοι πάντα ενισχυμένοι βγήκαμε από την κρίση και βγήκαμε από την κρίση όταν ανοίξα, ανοιχτήκαμε προς τον κόσμο και αξιοποιήσαμε τις παγκόσμιες ευκαιρίες και όχι όταν κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής και μετά ο κύριος Σέρκας. Ο κύριος Φεράτης. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι μόνο το 2011 προβλέπεται να σταθεροποιηθεί η απασχόληση στις χώρες Ευρωζώνης. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Σας ρωτώ, μήπως θεωρείτε ότι πάνω απ' όλα στους τομείς της κατασκευής ε, μεταποιήσεω χαμηλή προστάμενη αξία, μήπω η αναργία γίνει διαθροτική. Διότι βλέποντα τι συνέπειε μια συνεχού καθυστερήση της εισόδου νέων στην αγορά εργασία, ίσω θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κοινωνικέ εντάσει. Δύσκολο να τις χειριστούμε, κυρίως σε κάποιες περιοχές. Μήπως θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμη μια πολιτική κατεπίγουσα για να αντιμετωπιστεί ένας τέτοιος κίνδυνος, τέτοιας φύσεως. Διότι διαφορετικά η εμπιστοσύνη για την οποία μιλάμε, οι δείκτες που δείχνουν έξοδα, ε, η εξοπιστία των δικτών που μας δείχνουν μια έξοδα την κρίση, ίσως να είναι λιγότερο αξιόπιστη. Ο κύριος Σέρτζιο Κοφεράτη και μετά ο κύριο Κίγκαλο. Ο κύριος Σέρκας, συγγνώμη, πρώτο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εγώ θα ήθελα να κρατήσω τις τελευταίες σκέψεις ότι δεν υπάρχει οικονομικός δετερμινισμός, οικονομική τελειολογία. Όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα λάβουμε τα επόμενα χρόνια. Και θα ήθελα ο Επίτροπος Οικονομικών Θεμάτων να μιλήσει για τους αυτόματους δείκτες που διαδραματίζουν και πολύ θετικό ρόλο στην Ισπανία, για παράδειγμα. Πέραν του κινδύνου που υπάρχει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, Βέβαια δεν είναι αυτή η πέτη για, τα, για τα, τις τεράστιες που έγιναν στα δημόσια οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Και πώς εξηγείται η αύξηση κατά 10% του δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Τα διδάγματα από την κρίση σε μια χώρα σαν την Ισπανία που βρέθηκε στον κατάλογο των κακών μαθητών ενώ πριν από λίγα χρόνια ήμασταν πρωταθλητέ στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, μα δημιουργεί θλίψη. Και το θέμα είναι να έχουμε και ποιοτική απασχόληση. Στην ε, Ισπανία είχαμε προσωρινό χαρακτήρα μόνο 33% εποχιακή απασχόληση. Γιατί καλό είναι να μιλάμε για περισσότερη απασχόληση, αλλά μας ενδιαφέρει η ποιοτική απασχόληση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει δυνατό κάτι τέτοιο. Ο κύριο Βίνκι Κόλτ και μετά η κυρία Ντανούτα Σλαβίτσα. Πρέπει να πω ότι όταν διάβασα την έκθεση ανησύχησα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες ήταν, είχαν την επισήμανση alert. Και φοβάμαι ότι δεν τολμούμε να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Οι αλλαγέ ε, έως και 15% στο ΑΕΠ, οι οποίε θα πρέπει να το πιστούν στο μέλλον, τι θα πρέπει να σημαίνουν οι αλλαγές αυτές. Και θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει πιο ενεργά για το ποιες δομές θα πρέπει να αλλάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να βοηθήσουν με τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν δικαιούς ε, φόρους, γιατί έχουμε ε, μεγάλα προβλήματα με την ε, αθέμητη φορολογία. Έχουμε πολλά προβλήματα με τους φορολογικούς παραδείσους, πολλά μέτρα που αγγίζουν μόνο τον επιφάνειο του προβλήματος, που δεν μας βοηθούν να εξέλθουμε από την κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζουμε. Και οι χώρες που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα, κυρίως στο Νότο, είναι οι χώρες που καλούνται να πληρώσουν μεγαλύτερα επιτόκια τώρα σε σχέση με τις άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης. Και θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί σε ό,τι αφορά τα ευρωομόλογα και να ε, ρίξει τα επιτόκια για τις χώρες αυτές. Διακόπτη η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, ξεπεράσατε τον χρόνο αγόρευσης. Η κυρία Ντανούτα Γιασλοβιέκα και ζητώ συγγνώμη από τους, τις επόμενους την κυρία Παπαδουλό κυρία Γκρούνη, τρεις γυναίκες, διότι δεν θα έχουμε το χρόνο να ακούσουμε τις ερωτήσεις τους, διότι ο Επίτροπος πρέπει να μας εγκαταλείψει και εξαντλήσαμε και το χρόνο μας. Η κυρία Γιασκοβιέκα. τελευταία παρέμβαση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σε ό,τι αφορά την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα δημόσιων οικονομικών, έχουμε την πρόταση για μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών εργασίας προκειμένου να αυξηθεί η αποσχολησιμότητα. Υπάρχουν κάποια προγράμματα για διευκόλυνση των νέων για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, οι νέες οικογένειες, οι οικογένειες ε, νέων θα ήθελαν μια μετάβαση, θα φοβούνται με την αλλαγή του μοντέλου. Έχουμε και το πρόγραμμα για το 50 συν, για την τη δεξιδότηση. Και τι γίνεται με τις νέες γενιές. Μιλήσατε για τη μετανάστευση. Συνήθως στη μετανα... αποφασίζουν να μεταναστεύσουν οι νέοι άνθρωποι. Δεν θα πρέπει να προβλέψουμε μηχανισμούς για να στηρίξουμε τις νέες γενιές στην χώρα μας, ώστε να μην παίρνουν των οματιών τους και να περιοδεύουν από χώρα σε χώρα προκειμένου να βρουν μια θέση εργασίας. Θα πρέπει να διδαχθούμε από την παρούσα κρίση και να φροντίσουμε για τις νέες γενιές και για την καλύτερη δημογραφική κατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπη, σε μια τελευταία σειρά απαντήσεων. Σας ευχαριστώ. Τα θέματα που ανακύπτουν όταν ασχολούμαστε με συζήτηση για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων κοινωνικής και συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν είναι ευρύτατα και δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα και να τα εξετάσουμε σε μία συνεδρίαση ή επευκαιρία μίας έκθεσης. Σίγουρα θα συζητηθούν και σε επόμενα συμβούλια και σε επόμενε συνεδριάσει και σε επόμενε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Κοφεράτη, πολιτική εκτάκτου ανάγκη Μα εφαρμόζεται μια πολιτική εκτάκτου ανάγκη. Εφαρμόζεται μια τέτοια πολιτική ε, για την υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματο που μα αρέσει λίγο ή πολύ, αλλά χωρί χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν υπάρχει και οικονομικό σύστημα. Και ακόμη υποφέρουμε γιατί δεν υπάρχει ακόμη αποκατάσταση των δανείων και των πιστώσεων. Και παρά την ανάκαμψη δεν υπάρχει ανάκαμψη του δανεισμού. Επίσης και από νομισματική άποψη είναι ασυνήθιστα αυτά τα επίπεδα, τα χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων. Και αν θυμηθούμε τις απαρχές της κρίσης, οι καταβολές της κρίσης πολλές φορές ε, βρίσκονται σε μια ελαττωματική εκτίμηση των αγορών των κινδύνων από πλευράς αγορών δεν στάθμισαν αρκετά τους κινδύνους οι χρηματοπιστωτικές αγορές και ανέλαβαν κινδύνους ε, που ήταν, ε, ξεπερνούσαν τα λογικά όρια. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε ακόμη εξασφαλίσει τις εγγύησεις ότι έχουμε ε, βρεθεί σε ένα σταθερό μονοπάτι ανάκαμψης. Γιατί εντάξει, καταφέραμε να ανακόψουμε την κατακόρυφη πτώση της οικονομίας και τα τελευταία τρίμηνα προσπαθήσαμε να τη σταθεροποιήσουμε σε μια ζώνη θετικής ανάπτυξης. Άλλες χώρες επέτυχαν αυτή τη θετική ανάπτυξη πιο γρήγορα, άλλες με αργότερους ρυθμούς. Πάντως, ε, συμφωνώ ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και παρά την ε, ανάπτυξη της οικονομίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φλέγον ζήτημα της ε, ανεργίας και της ανάγκης αναδιάρθρωσης σημαντικών κλάδων της οικονομίας. Και για να βρούμε λύσεις χρειαζόμαστε φιλόδοξες και τολμηρές πολιτικές. Αλλά έχουμε επίγνωση ότι η κατάσταση αυτή είναι τόσο ιδιάζουσα που απαιτεί κάποια συνήθιστα οικονομικά μέτρα που σίγουρα δεν μπορούν να, να παραταθούν επαόριστον. Συμφωνώ κύριε Σέρκας ότι το ζητούμενο είναι μια ποιοτική απασχόληση. Κάτι όμως, κάτι τέτοιο προϋποθέτει μια οικονομία που θα επενδύει, που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, που θα είναι παραγωγική, που θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Χωρίς εύρωστη οικονομία δεν νοείται ποιοτική απασχόληση. Μπορεί να έχουμε κάποιες θέσεις εργασίας για κάποιο διάστημα, αλλά όχι ποιοτική απασχόληση. Και από την άποψη της σταθερότητας και από την άποψη της ικανότητας παράταση και στο μέλλον της θετικής κατάστασης και της ικανοποίησης των προσδοκιών των εργαζομένων. Θέλουμε υγιή οικονομική πολιτική για ποιοτική απασχόληση. Γιατί ποιοτική απασχόληση δεν νοείται χωρίς υγιή οικονομία. Παρόλο που δεν μπορούν όλες οι υγιείς οικονομίες να εξασφαλίσουν ποιοτική απασχόληση. Επίσης τώρα με το παιχνίδι αυτό των αυτόματων σταθεροποιητών. Όλοι προτιμούμε να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι που θα μας ωφελήσει όλους. Θα πρέπει να γίνουν σίγουρα κάποιες φορολογικές αλλαγές, αναφυσβήτητο κάτι τέτοιο. Και τώρα ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Σε ορισμένες χώρες εξετάζεται ο φόρος του άνθρακα σε άλλες χώρες αυξάνεται η φορολογία παρόλο που η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται. Γιατί καμία κυβέρνηση πριν από μερικά, από μερικά χρόνια θα τολμούσε να εξαγγείλει προγραμματικά την αύξηση των φόρων, την αύξηση φορολογίας. Αλλά χρειαζόμαστε ε, χρειαζόμαστε κρατικά έσοδα, γιατί εξαφανίστηκαν πολλά τέτοια έσοδα από την κρίση και χρειάζεται μία ανάκτησή τους. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα έχουμε προβλήματα για τη συζήτηση τη φορολογική. Και ο Λάσλο Κόβατς ε, μπορεί να σας, λέει, πει τι προβλήματα έχουμε στο ΕΚΟΦΗΝ. Αλλά χθες ήρθε και το τελευταίο κόλλημα για την κύρωση της συνθήκης Λισαβόνας. Αλλά ούτε και η συνθήκη της Λισαβόνας ε, έτυχε ομόφωνης ε, συνένεσης για τα φορολογικά και συζητήσεις ε, που και αποφάσεις που απαιτούν ομοφωνία θα γίνουν πολύ δύσκολα μεταξύ 27 χωρών μελών. Και η φορολογία είναι ένα από τα θέματα που απαιτεί ομοφωνία. Γι' αυτό και θα είναι δύσκολο να υπάρξει συνένεση σε επίπεδο 27 χωρών. Πάντως η συζήτηση γίνεται όλο και πιο πλούσια, πιο ενδιαφέρουσα. Μετά την ε, Λισαβόνα και μετά την κρίση παρά από ό,τι πριν σε ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων. Μακάρι να μπορούσα σε μισό λεπτό να βρω την μαγική φόρμουλα και το μαγικό ραβδί για να βελτιώσουμε την κατάσταση απασχόλησης και να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας στους νέους. Αλλά πιστεύω ότι οι νέοι θα εξασφαλίσουν καλύτερη θέση εργασίας ανάλογα με την παιδεία που θα λαμβάνουν. Όσο καλύτερη είναι η παιδεία και το επίπεδο της μόρφωσής του, τόσο καλύτερη απασχόληση θα βρουν. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Σίγουρα... Νομίζω ήταν πολύ πλούσια η ανταλλαγή των απόψεων. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ του διερμηνείς που συνόδευσαν μέχρι το τέλο των εργασιών μα. Αύριο θα τα ξαναπούμε σε 9.30 και όχι σε 9 το πρωί, 9.30 υπό την ηγεσία της Ελίζα Μπεθλίν που την ευχαριστώ που δέχτηκε να προεδρεύσει τον εργασιό μας. Καλό βράδυ και ζητώ συγγνώμη από τους τρεις συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να πάρουν το λόγο στη συζήτηση αλλά πρέπει να καταλάβετε πόσο περιορισμένη